So to start the meeting. Um, Αρχίζουμε τη συνεδρίαση. Έχουμε καλέσει τον ε, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Λίβιου Ντράγνεα, υπεύθυνο για την περιφερειακή ανάπτυξη και δημόσια διοίκηση. Και μαζί του είναι ο κύριος Ευγένιος Ορλάνδος Τεοντόροβιτς που είναι Υπουργός Ενωσιακών Πόρων. Θα αρχίσει ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ορίστε κύριε Αντιπρόεδρε. Θα μιλήσω στην Ρουμανική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκλησή σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που παρευρίσκομαι μπροστά σας σήμερα για να σας μιλήσω για ένα από, τους σπουδαιότερους στόχους της ρουμανικής κυβέρνησης και της δικής μου θητείας, δηλαδή την περιφερειακή αναδιοργάνωση της Ρουμανίας θα ήθελα να σας πω από την αρχή ότι η Ρουμανία βλέπει με πολύ ρεαλισμό το μέλλον της δημοσιονομίας στην Ευρώπη. Και γι' αυτό είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για το 2014. Και η αποφασιστικότητά μας φαίνεται από το γεγονός ότι όλον αυτόν τον χρόνο θα εφαρμόσουμε βαθύτατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τελικό μέχρι το τέλος του έτους να λήξει και αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί. Θα δημιουργηθούν νέες διοικητικές περιφέρειες για να είναι πιο καλά προετοιμασμένη η Ρουμανία να απορροφήσει ενωσιακούς πόρους κατά την, το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. πολδήμα. Οι τωρινές περιφέρειες έχουν μάλλον στατιστικό καθαρά χαρακτήρα και δεν έχουν περιφερειακή ταυτότητα χαρακτήρα και δικαιοδοσίες λήψης αποφάσεων. Και φάνηκε ότι δεν ήταν δυνατόν να διαχειριστούν σχέδια, προγράμματα. Οι περιφέρειες λοιπόν αυτές δεν μπορούν να διασφαλίσουν στις τοπικές κοινότητες δημοκρατική εκπροσώπηση. Είναι απλώς ένα σύστημα παρόμοιο με εκείνο των κομιτιών. Και αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στον στόχο της επίτευξης της ισορροπημένης ε, ανάπτυξης της χώρας. Από τότε που καθορίστηκαν αυτές οι λεγόμενες αναπτυξιακές περιφέρειες, το χάσμα μεταξύ αναπτυξιακού επίπεδου, ε, στα αναπτυξιακό επίπεδου μεταξύ τους έχει χειροτερέψει. Και σήμερα η Ρουμανία έχει μόνο μία πράγματι αναπτυγμένη περιφέρεια, εκεί όπου βρίσκεται το Βουκουρέστι. Όλες οι άλλες βρίσκονται σε πολύ χαμηλό αναπτυξιακό επίπεδο. Άλλο επιχείρημα για την υπέρ της αλλαγής του συστήματος είναι ότι οι περιφερειακές υπηρεσίες είναι μη κυβερνητικές, δεν ανήκουν στην κυβέρνηση και γι' αυτό δεν μπορούν να αρθούν στο ύψος της επίτευξης του στόχου της περιφερειακής ανάπτυξης. Έχουμε όμως 41 κομιτείες που είναι αρκετά μικρές διοικητικές μονάδες και γι' αυτό το τωρινό μας σύστημα καθώς και το σύστημα έγκρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων έχει δημιουργήσει πολύ κατακαιρματισμό και άχρηστο ανταγωνισμό μάλλον παρά συνεργασία. Έχουμε πολύ λίγη συνοχή λοιπόν περιφερειακά. Οι κομιτείες της Ρουμανίας όπως σας είπα είναι μικρές και άρα γνωρίζουν τις ανάγκες αλλά είναι υπερβολικά μικρές για να μπορέσουν να διαχειριστούν σοβαρά περιφερειακά προγράμματα. Από την άλλη η κεντρική κυβέρνηση έχει το όραμα να εφαρμόσει προγράμματα αλλά είναι πολύ μακριά από τις τοπικές κοινότητες και γι' αυτό υπάρχει αυτό το χάσμα στην ανάπτυξή μας. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται και ένα ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των τοπικών κοινοτήτων. Αρκετά κοντά σε αυτές για να γνωρίζει τα προβλήματά τους αλλά και αρκετά ψηλά ώστε να έχει ένα γενικότερο αναπτυξιακό όραμα και πρόγραμμα. Η γραφειοκρατία είναι υψηλή και γι' αυτό η περιφερειοποίηση πρέπει να συνοδευτεί και από αποκέντρωση ώστε να κατεβούν οι δικαιοδοσίες πιο κοντά στον κόσμο και τις τοπικές αρχές. Πρόθεσή μας είναι να τους δώσουμε αρκετές δικαιοδοσίες στις τοπικές αρχές ώστε να μπορούν να διαχειριστούν αυτά, αυτές τις νέες περιφέρειες και να χορηγούν ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες. Σε συμφωνία βέβαια και με τη στρατηγική του 2020 και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον με βάση αυτές τις νέες διοικητικές μονάδες και ενότητες που θα δημιουργήσουμε. Τις διοικητικές περιφέρειες δηλαδή, όχι <clears throat> πια τις αναπτυξιακές. Αυτές οι αλλαγές απαιτούν βέβαια προκαταρκτικά μια σωστή ανάλυση της κατάστασης στη Ρουμανία που γίνεται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση. Προσπαθούμε να την κάνουμε πολύ λεπτομερός ώστε να διαχειριστούμε καλύτερα τις μελλοντικές επαρχίες για να μπορούμε να εφαρμόσουμε πραγματική πολιτική συνοχή. Αυτό που θέλω να σας πω ως Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ότι η Ρουμανία έχει την ικανότητα να μαθαίνει από το παρελθόν της και γι' αυτό θα θέλαμε η αλλαγή να γίνει δίκαια και αποτελεσματικά και να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Και να είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα που θα αρχίσει από τον 1η Ιανουαρίου 2014, αγώνα απορρόφησης ενωσιακών όρων. Η αποκέντρωση βέβαια δεν είναι αυτός σκοπός, δεν το κάνουμε έτσι. Γιατί τελικός μας στόχος είναι να έχουμε λειτουργικές δομές με καλή διαχείριση που να μετατρέψουν τη Ρουμανία σε μια ισορροπημένη και αναπτυγμένη χώρα και που θα δώσει στους πολίτες την πρόσβαση σε καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Ως προσθέτης δικαιοδοσίες που θα χορηγήσει η κυβέρνηση στις τοπικές αρχές, στις νέες αυτές διοικητικές περιφέρειες, μεταξύ αυτών θα υπάρχουν τα υγειονομικά, η διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, κοινωνική προστασία, οικονομική ανάπτυξη, υποδομές, περιφερειακές υποδομές, τουρισμός, διοίκηση, γεωργία, προστασία του περιβάλλοντος, αντιμετώπιση επιγόντων περιστατικών, αθλητισμός, υψηλού επίπεδου μάλιστα. Γιατί θέλουμε να τελειώσουν όλα αυτά μέχρι το τέλος του έτους. Διότι προσπαθούμε να πετύχουμε υψηλό βαθμό απορρόφησης ενωσιακών πόρων και το σύστημα που έχουμε δεν δουλεύει καλά. Δεν θέλουμε λοιπόν να χάσουμε την ευκαιρία αυτή γιατί από τη μία είναι ο πρώτος χρόνος της διακυβέρνησής μας και άρα είναι η καλύτερη στιγμή για να ζητήσουμε και να δεχτεί ο κόσμος μεγάλες μεταρρυθμίσεις και από την άλλη η δυνατότητα να εφαρμοστεί αυτό το νέο σύστημα φέτος σημαίνει πριν αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Άρα προσπαθούμε να συνδυάσουμε την αναδιοργάνωση αυτή με τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης για το μελλοντικό πολιτικό. Αν δεν τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος του έτους θα χρειαστεί να περιμένουμε 7 ακόμη χρόνια. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε ότι οι Ευρωπαίοι θα δεχτούν στο επόμενο, στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο να μπορέσει η Ρουμανία να αλλάξει το διοικητικό της σύστημα δεύτερη φορά. Χρειαζόμαστε τις διοικητικές αυτές περιφέρειες επίσης για να μπορούμε να μπούμε στο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Δίκτυο και αυτό είναι νομίζω αναγκαίο γιατί έτσι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλύτερα με αυτό το δίκτυο. Η δε περιφερειοποίηση με την αποκέντρωση είναι διαδικασία που την περιμένουν πολλά χρόνια οι τοπικές αρχές στη Ρουμανία. Και δεν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να διεκπαιρεώσουν τα καθήκοντά τους όπως πρέπει. Είτε απευθυνθεί κανείς στον Δήμαρχο είτε στον Πρόεδρο ενό Δημοτικού Συμβουλίου, οι πολιτικοί εκεί δεν είναι σε θέση να τους βοηθήσουν γιατί δεν έχουν τη δικαιοδοσία να το κάνουν ούτε τα χρήματα η συγκέντρωση των δικαιοδοσιών στο Βουκουρέστι στην κεντρική κυβέρνηση είναι κακό πράγμα και τώρα χρειάζεται αποκέντρωση να μεταφερθούν εξουσίες και δικαιοδοσίες δηλαδή σε τοπικό επίπεδο και αυτή η διαδικασία θα απελευθερώσει πολλούς πόρους και δυναμικό δυνατότητες που μέχρι τώρα δεν τις έχουμε εκμεταλλευτεί. Όσο για τη συζήτηση για τη δημιουργία των περιφερειών και το χρονοδιάγραμμά της, η κυβέρνηση ενέκρινε ένα επίσημο χρονοδιάγραμμα για τη συζήτηση καταρχήν του προγράμματος Έχουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από μέλη ακαδημαϊκούς, καθηγητάς και άλλους Ρουμάνους και ξένους εμπειρογνώμονες εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Το Υπουργείο μου εξάλλου ασχολείται με, την, με όλα αυτά και έχει αναλάβει μία πολύ λεπτομερή μελέτη για να δει γιατί έχει τέτοια προβλήματα η Ρουμανία για την απορρόφηση των ενωσιακών κονδυλίων. Γιατί έχει αποτύχει στους στόχους που είχε καθορίσει από το 7 ήδη. Επίσης εξετάζουμε τους ακριβείς λόγους για τη δημιουργία της κάθε περιφέρειας και τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε τέτοια περιφέρεια για να δημιουργηθεί. Η περιφερειοποίηση δεν θα βασίζεται σε πολιτικά κριτήρια. Ούτε εθνοτικά. Το βασικό κριτήριο θα είναι λειτουργικό. Και όσα κριτήρια ταυτιστούν θα μπουν σε ένα μαθηματικό μοντέλο που θα μπορούν να το γνωρίσουν όλοι οι πολίτες ως σχέδιο που θα βασίζεται σε ακριβή ανάλυση. Αυτά δεν τα κάνουμε για ένα-δυο χρόνια, ούτε πρόκειται για καθαρά κομματικό θέμα. Είναι θέμα που αφορά τη χώρα ολόκληρη και θα δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ζήσουν καλύτερα στη χώρα τους. Επίσης θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι θα έχουμε μόνιμες επαφές με τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων διότι νομίζουμε ότι είναι σημαντικό οι εκπρόσωποι της Ένωσης να γνωρίζουν σωστά τις προθέσεις και τις προσπάθειές μας. Έχω ζητήσει και λάβει τη βοήθεια πολλών από σας που έχουν μεγάλη εμπειρία ως προς την περιφερειακή ανάπτυξη και καταλήγοντας θα ήθελα να σας μεταφέρω το μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να συμπληρώσουμε τη διαδικασία αυτή στα τέλη του, μέχρι τα τέλη του 2013 και αυτό προς όφελος των πολιτών και της χώρας ως πλήρως μέλους της Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε ε, κύριε Διπρόεδρε. Εμείς ε, ε, Λέμε πάντα την πρόεδρο τη κυβέρνηση. Ε, τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Τοντεροβίτση για τα εισαγωγικά σχόλια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι εξωτικά μέρη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή να έχουμε ανταλλαγή απόψεων για τα τρέχοντα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή τη ε, Ρουμανία ε, για τα διεθνωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχή. Για την ρουμανική κυβέρνηση είναι προτεραιότητα η απορρόφηση των ε, ταμείων και με τον στόχο αυτό Βουρκείο ε, Ενωσιακών Πόρων δημιουργήθηκε πέρσι το Δεκέμβριο και έχει στόχο να εφαρμόσει ένα πιο άμεσο συντονισμό των διάφορων επιχειρησιακών προγραμμάτων ε, μέσω μιας σχέσης με τις αρμόδιες αρχές και των διάμεσων φορέων. Ναι. Έχουμε δημιουργήσει ειδικά θέματα για κάθε πρόγραμμα προκειμένου να συνεργαστούμε στενά με τις αρμόδιες αρχές για να προωθήσουμε την εφαρμογή των προγραμμάτων από το επίπεδο του δικαιούχου και να αναλάβουμε στις δράσεις στο να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε δυσκολίες στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Επιπρόσθετα, ε, το μόνιμο καθήκον του Υπουργείου είναι να συγκεντρώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο εσωτερικό της Ρουμανικής Διοίκησης που μπορούν να συνεισφέρουν σε ένα επιτυχημένο ρυθμό απορρόφησης στην επόμενη κριτική κρίσιμη περίοδο και να αντιμετωπίσουμε το θέμα της χρηματοδότησης, την αύξηση της, απλούστευσης, της απλούστευσης αλλά και την ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου από τη Σκοπιά ε, του οριζόντιου συντονισμού ξεκίνησα στην συνεργασία με τον Υπουργό Δημοσίων Οικονομικών καθώς και με τα κύρια εθνικά ιδρύματα που έχουν να κάνουν με τις δημόσιες συμβάσεις. Η ικανότητα σε χρηματοδότησης ε, έχει θυχθεί από ε, διακεκομένες πληρωμές, όμως ελήφθησαν μέτρα για τη σημερινή προγραμματική περίοδο που αποτελούνται που μάλλον θέλουν να υποστηρίξουν τις εσωτερικές πληρωμές ε, για project ε, που εμπίπτουν ε, στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η Ρουμανία έχει βιώσει δυσκολίες στις δημόσιες συμβάσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Οι διαδικασίες οδήγησαν να έχουμε τρία προγράμματα σε προ-αναστολή από το 2009 στο 2011 και παρόλα αυτά λόγω των μέτρων που ελήφθησαν έχει γίνει σημαντική πρόοδος στο σχέδιο δράσης που συμφωνήσαμε με την Κομισιόν. Στο δεύτερο μάλλον στις αρχές του 2012 έχει εφαρμοστεί και έχουν ε, ληφθεί εκτατικές, εκτατημένες δράσεις. Ε, οι αρχές που είναι αρμόδιες για τις δημόσιες συμβάσεις ε, και η Εθνική Αρχή για την παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων και η αρχή που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έχουν αξιολογηθεί από τις ελεκτικές αρχές ελήφθησαν μέτρα για την παγίωση του ρόλου ελέγχου των διευθυντικών αρχών και υλοποιήθηκαν επαληθεύσεις δυνάμει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μηχανισμός για αυτή τη διοργανική συνεργασία μεταξύ των διευθυντών των αρχών και ε, των αρμοδίων αρχών για τις δημόσιες συμβάσεις ε, ενδυναμώθηκαν και έγιναν σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι έχουμε παληθεύσεις πιο συγκεκριμένες. Ε, το ε, θετικό ε, αποτέλεσμα αυτών των μέτρων φαίνεται ήδη και υπάρχει βελτίωση που μπορεί να φανεί σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης των διαγωνισμών και την τεκμηρίωση για την επίλυση των ε, προβλημάτων δημοσίου συμβάσεων δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων, της επίλυσης σύγκρουσης συμφερόντων συστηματικά. Η ρωμανική νομοθεσία περιλαμβάνει εκτατικές διατάξεις ε, που καθορίζουν ε, τον εντοπισμό της σύγκρουσης συμφερόντος καθώς ε, και μέτρα επιβολής κυρώσεων. Τα συγκεκριμένα βήματα που ελήφθησαν πέρσι προς την κατεύθυνση αυτή μας δείχνουν την πλήρη δέσμευση των ρουμανικών αρχών να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του νομικού, στάμενου νομικού πλαισίου και σε διαδικαστικό και σε επίπεδο ένας μηχανισμός αξιολόγησης εκπόστ έχει συσταθεί στο επίπεδο των αρχών διαχείρισης βάσει ε, της αξιολόγησης κινδύνου για να μπορέσει να εντοπιστεί, ε, να μπορέσει να εντοπιστούν πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Και τις επόμενες ε, δύο εβδομάδες θα στείλουμε και πρόσθετες πληροφορίες ε, για το θέμα αυτό, προκειμένου να επιληθεί το ζήτημα που αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και το μηχανισμό ελέγχου εξάντε ελήφθησαν πρόσφατα μέτρα για να ενδυναμωθεί η προ σύγκρουση συμφερόντων στις δημόσιες συμβάσεις μέσω της εξάντε επαλήθευσης στη συμφωνία με την Κομισιόν η Ρουμανία έχει ξεκινήσει μια διαδικασία πριν τον Οκτώβριο του 2012. Προγράμματα που αφορούν την ορθή διεξαγωγή των δημοσίων συμβάσεων, η Κομισιόν δέχτηκε το επίπεδο τη σχέση που προτείνεται από την Κομισιόν. Τώρα είμαστε σε ένα σημείο που υποβάλαμε έκθεση στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Φεβρουάριο για όλες τις αναπομείνασες ε, δράσεις. Έχουν ε, ληφθεί μέτρα σε οριζόντιο επίπεδο αλλά και για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τα προγράμματα η Κομισιόν θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει λάβει η χώρα. Ο Υπουργό ε, Ευρωπαϊκών Πόρων επίσης ε, αξιολογεί τη δυνατότητα πρόσβασης ε, στους ενωσιακούς πόρους για την επόμενη προγραμματική περίοδο, καθορίζοντας διάφορες στρατηγικές και καθορίζοντας το πλαίσιο σύμπραξης. Ε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκπόνησης της Συμφωνίας Σύμπραξης με σημαντικές ορμάδες εργασίας που έχουν συσταθεί σε επίπεδο Υπουργείων. Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται σήμερα στο να ολοκληρωθούν οι λεπτομέρειες και να εντοπιστούν οι προτεραιότητες σύμφωνα με το έγγραφο θέση της Κομισιόν, αλλά αντικατοπτρίζονται και συγκεκριμένες ε, αναπτυξιακές ανάγκες της Ρουμανίας. Ε, μία ευρεία εταιρική σχέση έχει δημιουργηθεί με τη δημιουργία της Θεσμικής Επιτροπής ε, για την Συμφωνία εταιρική σχέση από πέρσι τον Αύγουστο και άλλες 12 συμβουλευτικές επιτροπές και ομάδες τομεακές έχουν συσταθεί προκειμένου να εντοπίσουν οι κύριοι stakeholders να συμμετέχουν στην διαδικασία μια διαφανή προσέγγιση για την επιλογή των μελών αυτών των επιτροπών έχει εφαρμοστεί και πιστεύουμε ότι οι νέε απαιτήσει ε, για την εταιρική σχέση δεν ε, θα ε, επιφέρουν προβλήματα για τη Ρουμανία. Έχουμε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο υλοποιήσει διάφορες ε, συζητήσεις ε, για την εξάντε ερεσιμότητα. Επίσης, ε, το Υπουργείο Νοσιακών θα τεθεί μάλλον θα αρχίσει να λειτουργεί αφού σε επίπεδο κυβέρνησης θα έχει συζητηθεί η αιρεσιμότητα εξάντων. Ο μηχανισμός αυτός επίσης θέλει να διασφαλίσει την καλή εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων θα αξιολογήσουμε την ε, εφαρμογή ε, των προγραμμάτων σε διάφορα επίπεδα στη Ρουμανία και είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρίνηση. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Καταρχήν ο κύριος Λουγάν. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καθότι έχω γενέθλια σήμερα θα είμαι ε, ευγενικός απέναντι στους καλεσμένους μας. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκτιμούμε την παρουσία σας εδώ. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στους Ευρωπαίους νομοθέτες και τη Ρουμανική κυβέρνηση, άσχετα από το κόμμα από το οποίο προέρχονται. Και πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε κοινό μέτωπο όσον αφορά την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. Μπορώ να σας πω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε όλα τα λάθη και τις δυσκολίες ε, που ε, υπάρχουν στην ε, ρουμανική πολιτική αρένα και να βρούμε κοινέ λύσεις και υπάρχουν κάποια προβλήματα που συνδέονται με το παρόν πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το προσεχές το οποίο συζητιέται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αυτή τη στιγμή και έχω τρεις ερωτήσεις. Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά τρεις θα θέσω, πολύ συγκεκριμένες. Η πρώτη αναφέρεται στον κανόνα νη Η απόφαση του ε, Συμβουλίου, δηλαδή 7 και 8 ε, Φεβρουαρίου, ε, όπου ζητείται εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν για τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, το οποίο σημαίνει 4,5 ή 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ όσον αφορά την απορρόφηση. Οι λόγοι είναι γνωστοί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα το πρωί είχαμε συζήτηση με τον Επίτροπο Χάν. Την ίδια ερώτηση έθεσα και ρώτησα τον Επίτροπο ποια θα είναι η προσέγγιση της Κομισιόν για τις δύο χώρες αυτές που ζήτησαν παρέκκληση φαίνεται να μην υπάρχει συνένεση εντός της Κομισιόν. Ο Επίτροπος μας είπε ότι μόνο αυτός υποστηρίζει το αίτημα των δύο χωρών. Όλοι οι άλλοι επίτροποι είναι κατά. Συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν, η ρουμανική κυβέρνηση τι θα κάνει για να ε, ε, πετύχει αυτή την παρέκκληση, να περάσει από τον ΙΣΙΝ 2 στον ΙΣΙΝ 3 για να έχει καλύτερη δυνατότητα απορρόφησης ευρωπαϊκών ε, πόρων. Δεύτερη τεχνική ερώτηση. Όταν γίνατε μέλη της κυβέρνησης, η Ρουμανία είχε ποσοστό απορρόφησης 7%. Δεδομένου ότι 70% κάλυπταν οι συμβάσεις μέσα σε ένα χρόνο έχετε αυξήσει το ποσοστό ε, απορρόφησης μόνο κατά 3,4%. Κατά τη γνώμη μας υπάρχει τεράστιο κενό ανάμεσα στο 78% ε, ως ε, ποσοστό που καλύπτουν οι συμβάσεις και, την, και αυτά που έχει πετύχει η κυβέρνηση μέσα σε ένα χρόνο όσον αφορά το επίπεδο απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων. Τέλος, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας ε, είναι η συμφωνία με το Διεθνές Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Υπάρχει μια σειρά συγκεκριμένων θεμάτων, όπως είναι η αύξηση της ε, συγχρηματοδότησης από 85% σε 90% για τα περιφερειακά ταμεία και ε, να φτάσει το 100% για τη, για γεωργική ανάπτυξη. Δεν μιλάμε λοιπόν για νέα δανειακή σύμβαση, θα θέλαμε όμως να γνωρίζουμε αν η παρούσα κυβέρνηση θα συνάψει νέα συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια προληπτική συμφωνία, να το πούμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ, η Κωνσταντσε Κρέμερ. Ευχαριστώ πολύ πολλές ερωτήσεις. Ε, δεν ξέρω αν ε, υπάρχει ακόμα χώρος για μένα. Χάρηκα πολύ που άκουσα το φιλόδοξο πρόγραμμα της κυβέρνησής σας. Να δημιουργηθούν ε, νέες διοικητικές περιφέρειες. Δύο ερωτήσεις έχω. Θα πρέπει να ετοιμάσετε τη νέα περίοδο τώρα που κλείνει η πρώτη και θέλετε να αλλάξετε το σύνολο της, ε, της διάρθρωσης. Ε, τι θα γίνει λοιπόν ε, με τις περιφέρειες, με τα επιχειρησιακά προγράμματα σε σχέση με την δική μας ε, εικόνα που έχει αναφερθεί στον τριμερή διάλογο και την ε, αρχή της εταιρική σχέσης. Και η άλλη ερώτηση είναι ότι ουσιαστικά δημιουργείται μια νέα δομή, η οποία αν έχω καταλάβει σωστά, στόχο έχει την ε, ε, διαχείριση των ε, επιχειρησιακών προγραμμάτων πρόκειται για αποκέντρωση, αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι χρειάζεστε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι να έχουν σχετικές διοικητικές γνώσεις. Το δυναμικό αυτό λοιπόν πώς προβλέπετε να δημιουργηθεί και αρκεί, αρκούν αυτά που μπορεί να δώσει η Κομισιόν ως οικονομική υποστήριξη. ώστε να, το νέο, ώστε να ξεκινήσει το νέο διάστημα με, ε, με επακές δυναμικό και με καλό τρόπο. Ε, η Κορνέλια Έρνστ και κατόπιν να ζητήσουμε από τους υπουργούς να απαντήσουν. Ναι, ευχαριστώ πολύ. από την παρουσίασή σας. Ε, καταλαβαίνουμε ότι η Ρουμανία ε, βρίσκεται μέσω μεγάλων αλλαγών ε, και, στην, και στον διοικητικό τομέα, κάτι που συνδέεται και με την δημοκρατία. Τα γνωρίζουμε αυτά και στην Ανατολική Γερμανία τα έχουμε δει αυτά. Γνωρίζουμε λοιπόν τα προβλήματα που προκύπτουν. Και η πρώτη μου ερώτηση είναι στις αλλαγές αυτές στον διοικητικό τομέα που έχουν σημαντικές ε, συνέπειες ε, για τις περιφέρειες, σε τι υποστήριξη χρειάζεστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως χρειάζεστε βοήθεια από χώρες με παρόμοια δομή. Αυτό θα ήταν σημαντικό. Μήπως μπορείτε κάτι να πείτε γι' αυτό. Δεύτερον, είχατε μια σειρά δυσκολιών όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση. Πιστεύετε ότι μπορούν να λυθούν τα προβλήματα στο προσεχές χρονικό διάστημα. Ε, τι έχετε κάνει εκεί όσον αφορά τις ε, σχετικές βελτιώσεις και ξέρετε ότι έχουμε μεγάλες συζητήσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ότι το Κοινοβούλιο ε, είναι κατά. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ε, εσείς πώς βλέπετε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και αν μπορείτε να μας πείτε κάτι σχετικά με τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να σχολιάσετε τώρα? Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ίσως ε, και ο υπουργό Πετροβίτης θα απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις σε ό,τι αφορά τον κανόνα νησυντρία. Και η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Ρουμανίας θα πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε η υπόσχεση που δόθηκε και στη Ρουμανία και στην Σλοβακία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να τηρηθεί. Θέλουμε οι εμπειρογνώμονες της Κομισιόν να βρουν ένα τεχνικό τρόπο για να εκπληρωθεί αυτή η υπόσχεση. Δεν πιστεύουμε ότι η μελλοντική αλλαγή, η μελλοντική τροποποίηση στον κανονισμό είναι δυνατή γιατί αυτή ήταν μια πολιτική απόφαση υψηλού και συνεχίζουμε να καταβάλουμε προσπάθειες. Πολύ σύντομα θα συναντηθούμε με την Επιτροπό Χάν και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό, θα συνεχίσουμε να ζητάμε την υποστήριξή του για να επιλύσουμε αυτό το θέμα και να βρούμε μια καλύτερη λύση. Όμως, όπως και να έχει, η Ρουμανία πρέπει να συνεχίσει με την εφαρμογή όλων των δράσεων που έχουμε αποφασίσει, έτσι ώστε η βαθμός απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων να αυξηθεί. Σε ό,τι αφορά την ε, πιθανή νέα συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Τομείο του Παγκόσμια Τράπεζα και την Κομισιόν είναι η πρόθεσή μας να υπογράψουμε μια τέτοια προληπτική συμφωνία, όχι απαραίτητα επειδή χρειαζόμαστε χρήματα, αλλά οι διαπραγματεύσεις με αυτούς τους τρεις εταίρους έλαβαν χώρα τον Ιανουάριο. Έχει καταρτιστεί μια επιστολή προθέσεων, ε, μέσα της οποίας ε, η Ρουμανία έχει κάνει ρεαλιστικές δεσμεύσεις που είναι απολύτως απαραίτητες για τη Ρουμανία. Και κάναμε αυτές τις δεσμεύσεις όχι για να απαντήσουμε στο Διεθνές Μεσοδοτικό Αμείο και στις απαιτήσει του και στις απαιτήσει της Κομισιόν, αλλά επειδή χρειαζόμαστε την υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων. Εμεί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για τη Ρουμανία να έχει μια τέτοια συμφωνία με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γιατί αυτό μας δίνει μια πρόσθετη αξιοπιστία και μας βοηθά να έχουμε καλύτερες συνθήκες όταν δανειζόμαστε χρήματα από τις ε, ιδιωτικές αγορές. Αλλά επίσης ε, πρέπει να προβούμε και στην αναδιάρθρωση που χρειάζεται η Ρουμανία σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις ε, της κυρίας κρεμ. Μπορώ να πω ότι ο αριθμός πυρογνωμόνων που είναι απαραίτητος για να λειτουργούν ε, καλά στο μέλλον οι διοικητικές ε, περιοχές, τα διοικητικά μετά, δεν είναι και τόσο υψηλό. Έχει η Ρουμανία αυτούς τους εμπειρογνώμονε αυτή τη στιγμή. Εργάζονται στις υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης, που αυτή τη στιγμή λειτουργούν ως ενδιάμεσα ιδρύματα, ως ενδιάμεση φορείς. Επομένω, υπάρχουν αυτοί οι προγνωμόνε, υπάρχουν οι δομές και βέβαια αυτό το είχαμε κατά νου όταν αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτές τις διοικητικές περιφέρειες. Και φυσικά αυτές οι δομές θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη και υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα την αρχιτεκτονική των επιχειρησιακών προγραμμάτων, νομίζω ότι η κυβέρνηση θα θέσει τις τελικές ε, πινελιές ε, στην πρόταση τις επόμενες ημέρες και κατόπιν θα στείλουμε την πρόταση της Κομισιόν, στην Κομισιόν, με συγχωρείτε, η περιφέρειες θα έχουν αρμοδιότητες ε, διαχειριστικών αρχών και ελπίζουμε να μπορέσουμε να πείσουμε την Κομισιόν να δεχτεί αυτή τη λύση, έτσι ώστε το 2014, το 2015 και ίσως και το 2016 οι δομές αυτές καθώς θα έχουν αναπτύξει τις διοικητικές τους ικανότητες, να μετατραπούν σε κανονικές διευθύνουσες αρχές. Θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί κατά τη δικασία αυτή για να μην θέσουμε ποτέ σε κινδύνο την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επίσης, όπως σας είπα, ήδη οι φορείς απασχολούν υψηλά εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες και εμείς έχουμε φτάσει σχεδόν και στο 100% των συμβάσεων στο δικό μου Υπουργείο και έχουμε για ένα καλό ποσοστό πρόφησης. Έτσι λοιπόν αυτές οι υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης ε, είναι στελεχωμένες με το κατάλληλο προσωπικό. Σε ό,τι αφορά τώρα την μεταρρύθμιση των ε, μελλοντικών διοικητικών περιφερειών στα πλαίσια της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης όλες οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τα Συμβούλια για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Κοινωνία των Πολιτών, ε, διάφορες ενώσεις, οι κοινωνικοί εταίροι, όλοι αυτοί θα είναι διαρκώς ενημερωμένοι για τη διαπραγματευτική διαδικασία έτσι ώστε την 1η Ιανουαρίου 2014 οι περισσότεροι εξ αυτό θα πρέπει να έχουν έτοιμες τις αιτήσει τους για να μπορέσουν να ξεκινήσουν την απορρόφηση των κονδυλίων το συντομότερο και μόλις ξεκινήσει φυσικά το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα για να απαντήσω στην κυρία Έρνστ. Πράγματι, η αναδιάρθρωση της διοίκησης είναι μια δύσκολη διαδικασία και πολύπλοκη διαδικασία. Χρειαζόμαστε υποστήριξη και Έχουμε ήδη πολλές συζητήσεις με συναδέλφους από άλλα κράτη-μέλη, οι οποίοι δέχτηκαν να μας βοηθήσουν και ελπίζουμε ότι μετά τις 15 Απριλίου θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να οργανώνουμε σεμινάρια και εργαστήρια με εμπειρογνώμονες από άλλες χώρες. Και έχω κατά νου ανθρώπους από την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία που έχουν πάρα πολλή εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Χρειαζόμαστε αυτή την εμπειρογνωμοσύνη γιατί Κατά τη διάρκεια μια τόσο πολύπλοκη διαδικασία ε, πέρα από του κινδύνου που έχουμε ήδη σκεφτεί, μπορεί να ανακύψουν και άλλοι κίνδυνοι. Επομένω, δεν ε, θέλουμε να επενεφεύρουμε τον τροχό, απλώ θέλουμε να προσπαθήσουμε να μάθουμε από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και την εμπειρία του. Ό,τι αφορά τώρα τι τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης. Εμείς ε, σκοπεύουμε να εισαγάγουμε ένα μηχανισμό που θα αντικαταστήσει το μηχανισμό αποζημίωσης, αντιστάθμισης. Έτσι λοιπόν οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει πλέον να αναζητούν πόρους για να κάνουν μία πληρωμή εκ των προτέρων και κατόπιν να μας στείλουν την απόδειξη και να περιμένουν τα χρήματα, αλλά φυσικά θα πρέπει να στείλουν τα, τα απαραίτητα έγγραφα, θα ελέγξουμε τα έγγραφα, θα τους πληρώσουμε και σε λίγες μέρες οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν τα χρήματα οι τοπικές αρχές ε, δεν χρειάζεται πλέον να ζητούν χρήματα αλλού προκειμένου να καλύψουν ε, αυτή την περίοδο για να αποφασιστεί η εκταμίευση. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο γιατί ο κύριος στόχος τον οποίο οι τοπικές αρχές δεν έχουν μπορέσει να βρουν επαρκή χρηματοδότηση είναι ακριβώς ότι πρέπει ε, εκ των προτέρων να βρουν τα κονδύλια και μετά να περιμένουν την εκταμίευση, την αποζημίωση. Οι συνάδελφοι από το Υπουργείο Οικονομικών διερεύνησαν τη δυνατότητα να συμμετάσχει και το τραπεζικό σύστημα στη χρηματοδότηση αυτών των project. Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει. Αν σταθούν με επιτυχία, θα μπορούσαμε να έχουμε έγκαιρα οικονομικούς πόρους, έτσι ώστε να άρουμε την πίεση από τις τοπικές αρχές. Και επίσης, ξεκινήσαμε μια διαδικασία μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης. Ε, μιλάμε και για μεταρρύθμιση του σε σχέση με το να έχουμε ξεκάθαρους κανόνες για τα πρότυπα του κόστους. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους και τα εναπομείνατα ποσά να τα κατανείμουμε για την ενδυνάμωση ε, του προϋπολογισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επομένως, ε, όσα κονδύλια δεν έχουν επενδύσει σήμερα θα πάνε προς τη χρηματοδότηση. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την απόφαση του Κοινοβουλίου. Για μας είναι πολύ ευνοϊκή η απόφαση αυτή και σκέφτομαι τη δυνατότητα ευελιξίας εντός ε, του δημοσιονομικού εγχειρήματο. Μας αρέσει αυτή η ιδέα της ευελιξίας και ελπίζουμε ότι ο τριμερής διάλογος θα στεφθεί με επιτυχία και ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί ο προπολογισμό ε, σε λογικό χρονικό διάστημα. Και ο κύριος Στεντροβίτση θα ήθελε να απαντήσει ορισμένε από αυτές τις ερωτήσεις. Να απαντήσω στο θέμα σχετικά με τον κανόνα νη συν 3. Έχουμε συζητήσεις με, ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τον μηχανισμό που θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε τον κανόνα νήσιν 3 στην Ρουμανία και την Σλοβακία. Από την άλλη καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε στο τέλος της χρονιάς να φτάσουμε το 6,5 δις ε, ε, όριο των ε, τιμολογίων. Ελπίζουμε λοιπόν να μπορέσουμε να κάνουμε τις πληρωμές ώστε να αποφευθεί η εφαρμογή του κανόνα. Από την άλλη συνομιλούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρούμε τρόπο να εφαρμόσουμε τον κανόνα νήσιν 3 στη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Όσον αφορά το ποσοστό που κάλυπταν οι συμβάσεις, 78% πέρσι, πιστεύω ότι εδώ πρέπει να έχουμε πιο ρεαλιστική προσέγγιση θα πρέπει να κοιτάξουμε τις συμβάσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, διότι ε, αυτό το ποσοστό, και, όχι το ποσοστό χρηματοδότησης, διότι αυτό είναι πιο ρεαλιστικό. Έχουμε 78% ε, ποσοστό για συμβάσεις όπου έχουμε υπογράψει με τους τελικούς δικαιούχους. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι η δημόσια σύμβαση αυτή καθ' αυτή, διότι αυτό μα ε, δίνει έναν υπολογισμό του επίπεδου πληρωμών. Είχαμε αύξηση περίπου 3% από την αρχή της χρονιάς και αυτό μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα μπορέσουμε να φτάσουμε ε, τον στόχο μας. Ε, έχουμε κάποια βασικά στοιχεία, απλοποίηση, αύξηση της διαφάνειας ε, σε όλη την διαδικασία Ευρωπαϊκών Ταμείων, ε, ε, μηδενική ανοχή όσον αφορά την σύγκρουση συμφερόντων, διαφθορά κλπ. Να διαχειριστούμε τις περιπτώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουμε και να διασφαλίσουμε αλλαγή στην οτροπία. Κάθε μέρος του συστήματος θα πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. και θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις που λαμβάνουν, διότι πολύ συχνά η έλλειψη απόφασης είναι χειρότερη από ε, οποιαδήποτε κακή απόφαση. Όσο θα προχωράει η διαδικασία, αυτό δεν θα σημαίνει απαραίτητα ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των ε, ανθρώπων που συμμετέχουν στο σύστημα. Όπως είπε ο αναπληρωτής ε, πρωθυπουργός, θα πρέπει να ε, βρούμε ισορροπία ανάμεσα στον αριθμό των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτές τις νέες μονάδες και την αποτελεσματικότητα των μονάδων. Και θα πρέπει βέβαια να σκεφτούμε το θέμα της κατάρτισης σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές. Πιστεύω ότι η υποστήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που ελπίζω θα συνεχίσει να παρέχει ε, είναι πολύ σημαντική. Μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στάθηκε στο πλευρό μας ε, όποτε χρειαστήκαμε βοήθεια και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Έχουμε συχνές επαφές πάνω στα θέματα αυτά. Και θα ήθελα να πω και λίγα λόγια σχετικά με τη, χρηματοδο... με συγχρηματοδότηση. Θα ήθελα να επιμείνω στην ανάγκη να μειωθεί το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην πληρωμή ενός τιμολογίου και τη στιγμή που ζητάμε επιστροφή του ποσού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να ε, μειωθεί ανάλογα και η δημοσιονομική προσπάθεια. Ε, στα μελλοντικά επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να έχουμε δημοσιονομικά προγράμματα ε, ώστε να μπορούμε να χρηματοδοτούμε και άλλα προβλήματα τα οποία θα, προγράμματα τα οποία θα ωφελήσουν και τους ανθρώπους και τις, και τις τοπικές αρχές. έτσι ώστε να ε, μην είναι τόσο μεγάλο το δημοσιονομικό άχθος. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω, όπως είπα και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, θα στείλουμε σχέδιο δράσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος της χρονιάς, που θα περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που προβλέπει η Ρουμανική Κυβέρνηση για το 2013 από τη μία για να ε, αυξήσουμε την απορρόφηση, να ε, ανακτήσουμε το χαμένο χρόνο και από την άλλη θα έχουμε και τα μέτρα που θα μας ε, ετοιμάσουν για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Πέτρου, μισό λεπτό σου δίνω και μην ξεχνάς ότι έχεις γενέθλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα για να ε, για να είμαστε σωστοί. Ο Υπουργός ε, αναφέρθηκε στην ε, στην μάλλον μικρή πιθανότητα να υιοθετηθεί η παρέκκληση. Ο Επίτροπος όμως είπε ότι είναι ανοιχτό απέναντι σε εναλλακτικέ λύσει για να μπορέσει η ρουμανική κυβέρνηση να απορροφήσει τους πόρους που δεν κατάφερε να απορροφήσει το τελευταίο χρόνο. Ε, ποια λοιπόν είναι τα εναλλακτικά μέτρα που προτείνετε για, τα, για να απορροφηθούν τα 4,5 με 5 δι. Ευχαριστώ. Ε, Καταρχήν, ε, χρόνια πολλά κύριε Λουχάν. Σε εύχομαι κάθε επιτυχία ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε πως η Κομισιόν θα βρει μια τεχνική λύση και την κατάλληλη νομοθετική λύση έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα νήσιν 3 αυτή την υπόσχεση μάλλον σχετικά με τον κανόνα νήσιν 3 εμείς ε, εργαζόμαστε επί εναλλακτικών λύσεων και θα παρουσιάσουμε τις λύσεις αυτές στον Επίτροπο Χάν Πρόεδρος ε, για να δούμε αν συμφωνούμε επί το του Συμβουλίου. Είναι πολύ ξεκάθαρα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου νήσιν 3 για όλους. Η Σλοβακία και η Ρουμανία αναφέρονται στο πλαίσιο της τρέχουσας περίοδου και ζητήθηκε από το Συμβούλιο, ζήτησε το Συμβούλιο από την Κομισιό να εξετάσει με ποιον τρόπο αποφεύγοντας οποιασδήποτε περικοπές για τη Σλοβακία και τη Ρουμανία για το ε, περίοδο 2007-2013 μπορεί να βρεθεί συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγή, του σημερινού κανονισμού. Έτσι λοιπόν υπάρχει έτοιμα να διερευνήσει η Κομισιόν κάθε πιθανό τρόπο για να αποφευχθεί η απώλεια κονδυλίων στη Σλοβακία και στη Ρουμανία στην τρέχουσα περίοδο και με τη δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού. Αυτό είπε το Συμβούλιο. Τώρα τι θα κάνει η Κομισιόν είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα, πέντε άτομα έχουν ζητήσει το λόγο και έχουμε δέκα λεπτά. Αν ξεπεράσετε το ένα λεπτό λοιπόν, μάλλον θα είναι δύσκολο να σας απαντήσουν ε, οι προσκεκλημένοι μας ε, Νίκο και μετά ο Βίκτορ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρο. Ε, Πρόεδρε. Ε, κατάλαβα ότι έχετε ένα καλή πρόθεση να κάνετε μεταρρύθμιση και να πάτε προς πιο περιφερειακή οργάνωση της χώρας και ταυτόχρονα όμως την ίδια περίοδο θα πρέπει να γίνει προετοιμασία. Και υπάρχει και ένα τρίτο θέμα ότι η μεταρρύθμιση του τρόπου που δουλεύει ένα κράτος δεν είναι απλώς η δημιουργία ορισμένων επιτροπών, αλλά η αλλαγή όλης της κουλτούρας, η στελέχωση των υπηρεσιών, η αναβάθμιση των ικανοτήτων των ανθρώπων που στην περιφέρεια θα πρέπει να αναλάβουν ρόλους και όλο αυτό να είναι δεμένο σε ένα σχέδιο. Αλλά από την άλλη μεριά κατάλαβα ότι ακόμα είσαι στην, στο επίπεδο της μελέτης. Δηλαδή, περιμένετε αποτελέσματα κάποιας μελέτης για να μπορέσετε να καταλήξετε στο πώς θα προχωρήσετε. Ε, φοβάμαι, επειδή έχω την εμπειρία από την Ελλάδα, ότι οι προθέσεις είναι πάντα καλές, αλλά στο τέλος η υλοποίηση των προθέσεων γίνεται με έναν τρόπο που λειτουργεί καταστροφικά. Δηλαδή, η μεταρρύθμιση στην Ελλάδα για τις περιφέρειες έγινε το 2010, αλλά ακόμα δεν έχουν αναλάβει αυτού του ρόλου του περιφερειακού σχεδιασμού. Και ε, αν δεν υπάρχει και μια στρατηγική, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και το δεύτερο δεν κατάλαβα, ακριβώ είπατε ότι όταν θα φέρουν οι δικαιούχοι τα τιμολόγια θα πληρώνονται. Αναφέρθηκε ότι οι τράπεζε θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη ε, δραστηριότητα, εφόσον το δεχτούν, αλλά εκεί θα προκύψει και ένα θέμα με ε, επιτόκια κλπ. και θα είναι από εθνικού πόρου, θα είναι από το τραπεζικό σύστημα και αν δεν δουλέψει το τραπεζικό σύστημα, ποια είναι η εναλλακτική λύση για να πληρώνονται γρήγορα οι δικαιούχοι όπως αναφέρατε πριν. Thank you. Thank you so much, Danuta. Ευχαριστώ, Δανούτα. Θα μιλήσω ρουμάνικα. Λοιπόν, ε, θα μιλήσω ρουμάνικα για δύο λόγους. Έχουμε δύο υπουργούς παρόντες στην Επιτροπή μας ε, σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ που ε, μια διατύπωση που φαίνεται να είναι απαγορευμένη στο Βουκουρέστι, η περιφερειακή μεταρρύθμιση, ε, ε, πια χρησιμοποιείται επίσημα στη χώρα μου. Αυτό προς όφελος και της Ευρώπης και της χώρας μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή. Δύο ερωτήσεις έχω. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιστήσει την προσοχή ε, της Ουρμανικής κυβέρνησης ε, στο θέμα της ε, καταπολέμησης της διαφθοράς και, της, και του μεγάλου κινδύνου για απάτη που υπάρχει. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση της Ρουμανίας αυτή τη στιγμή για να μειώσει τον κίνδυνο απάτης και δεύτερον πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει τις προσπάθειες ενός κράτους μέλους της Ρουμανίας δηλαδή να εφαρμόσει η περιφερειακή μεταρρύθμιση το 2013, διότι είναι πάρα πολύ απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο στη χώρα μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κατρίν Πέτρου. Μια πολύ σύντομη ερώτηση. Μιλήσαμε γι' αυτό σήμερα το πρωί και θα ήθελα να ακούσω τι σκέφτεστε εσείς για τη μικροοικονομική αιρεσιμότητα και πώς πιστεύετε ότι θα ενταχθεί αυτό στα δικά σας σχέδια. Ευχαριστώ. σα, Ματούλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους δύο αξιότιμους Ρουμάνους προσκεκλημένους μας. Εγώ έχω συνεργαστεί μαζί τους ε, το 2004 μέχρι το 2008 ως ε, πρόεδρος του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή με τον αντιπρόεδρο μας συγχωρείτε της κυβέρνησης, ε, τον ε, κύριο Ντράγκνε, συνεργαστή, αλλά και με τον κύριο Τεντροβίτσο, ο οποίος και τότε ήταν υπουργό. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε τις, την απορρόφηση των κονδυλίων στη Ρουμανία, πρέπει να συνεισφέρουμε στη συνολική οικονομική ανάπτυξη της Ρουμανίας. Εγώ έχω να κάνω κάποια σχόλια, μιλώντας για περιφερειοποίηση. Θα θέλαμε να σας συγχωρούμε Κύριε Αντιπρόεδρε, πράγματι πρόκειται για τεράστια ευθύνη, αλλά πρέπει να αναλάβετε δράση φέτος και μάλιστα πολύ γρήγορα, μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη όσα είπε και η συνάδελφος η κυρία Κρέλ. Τώρα προετοιμάζουμε τα έγγραφα για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και για τα επιχειρησιακά προγράμματα και θέλαμε ήδη να το κάνουμε από το 2012, αλλά θα το κάνουμε το 2013, αλλά δεδομένη της δικής σας ε, εμπειρίας, ε, κύριε Αντιπρόεδρε, ε, πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε και επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Γιατί θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα υπάρχουν ε, αρχές σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο κομιτείας. Στην ε, Ρουμανία έχουμε κομιτείες που έχουν ε, κάτω από 300.000 κατοίκους και υπάρχει μεγάλη επικάλυψη αρμοδιοτήτων σε αυτές τις συγκεκριμένε κομιτείες. Αυτό θα πρέπει να ληφθείτε όντως υπόψη. Αλλά και πάλι μιλώντας για τις περιφέρειες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχει δει λειτουργήσει ή οι υπηρεσίε περιφερειακή ανάπτυξη ε, λειτουργούν εδώ και καιρό και ίσως πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τα αποτελέσματά τους. Ε, πρέπει να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις για θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες ε, σε επίπεδο τοπικής ε, διοίκησης. Δηλαδή πώς γίνεται εκεί η εφαρμογή σε εκείνο το επίπεδο, γιατί εκεί έχουμε προβλήματα και εκεί δεν έχουμε εμπειρογνώμονες και αν τους έχουμε δεν μπορούμε να τους διατηρήσουμε στο σύστημα γιατί είναι ιδιαίτερα χαμηλόμισθοι και έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Οποιαδήποτε ομάδα ασχολείται με την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων έχει τεράστιε ευθύνε. Σε αυτά τα θέματα πρέπει να βρούμε λύσει, γιατί διαφορετικά θα μπορέσουμε ποτέ να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση. Και ελπίζω, κύριε Υπουργέ Τιοντοροβίτση, ότι θα μπορέσετε να τα καταφέρετε. Σας ε, ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε. Είναι προφανέ ότι ασχολείστε με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για πολλά χρόνια και ίσω μαζί με τον ε, κύριο Αντιπρόεδρο θα μπορέσετε να παρουσιάσετε συγκεκριμένα βήματα σε σχέση με την εφαρμογή. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα νέα μέτρα που έχετε κατά νου για να αυξηθεί το ποσοστό της απορρόφησης των κονδυλίων, όχι μόνο για σήμερα, αλλά και για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Δεν θέλω η Ρουμανία και πάλι να χάσει το τρένο όπως συνεβεί ήδη. Θα πρέπει να δούμε και τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση. Ο Επίτροπο Χάν μα είπε ότι την ήθελε τον Ιούνιο. Πρέπει να μελετήσουμε και το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Έχουμε Ε, κάνει κάποια βήματα, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη εξέλιξη. Ευχαριστώ, κυρία Ταντσίλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε ε, Αντιπρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Βλέπουμε ότι υπάρχει νέα προσέγγιση όσον αφορά τις σχέσεις ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή μας. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει νέα προσέγγιση στον τρόπο που ενημερώνουμε τους ε, συναδέλφους μας ε, από τα υπόλοιπα 26 κράτη-μέλη δεδομένης της ε, πρακτική προσέγγιση, τη ρεαλιστικής προσέγγιση σα ε, στην περιφερειακή πολιτική στην ε, Ρουμανία. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν προβλέπετε και συνέχεια της παρουσίας σας στην Επιτροπή αυτή, ώστε να αποτρέψετε παρερμηνία των τιμάτων που αναλαμβάνετε στη Ρουμανία. Χρειάζεται διαφάνεια θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο, στην στο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη Ρουμανική Κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου ε, να προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος όσον αφορά την ε, αναδιάρθρωση της ε, δημόσιας διοίκησης. Είναι πολύπλοκη η διαδικασία αυτή και μπορεί να μην ήμουν αρκετά σαφής κατά την πρώτη μου παρουσίαση. Δεν πρόκειται για μια επιφανειακή προσπάθεια, είναι κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια οι εκπρόσωποι των ε, δημοσίων θεσμικών οργάνων ε, έχουν εκπονήσει μελέτες οι οποίες έχουν ενοποιηθεί σε μια, ε, σε μια λεπτομερή ανάλυση σχετικά με το πού θα πρέπει να προχωρήσουμε στην αποκέντρωση, στην ανάθεση εξουσιών και ποια θα πρέπει να είναι η αρχιτεκτονική των διοικητικών περιφερειών στο μέλλον κλπ. Και ένα δεύτερο θέμα. Εάν στη Ρουμανία έχουμε δικαιούχο ενός προγράμματος, ο οποίος θέλει να λάβει χρήματα, θα πρέπει να καταβάλει τα χρήματα και κατόπιν να περιμένει την επιστροφή ε, των ευρωπαϊκών πόρων. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι ε, με βάση το τιμολόγιο που ε, λαμβάνει από τον ανάδοχο να ε, μεταφέρονται πιο γρήγορα τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να απαντήσω στον κύριο Ποσινάρου, ε, όλες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ρουμανία προέρχονται από κάποια σημαντικά λάθη. Όσον αφορά τα μέτρα που έχει αναλάβει η κυβέρνησή μας και που θα αναλάβουμε στο μέλλον, συμπεριλαμβάνουν και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής για να αποφύγουμε πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Ε, και το σύστημα αυτό ε, θα μας προειδοποιεί σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο να βοηθά τις ε, δημόσιες αρχές ε, να αποφύγουν ε, τη σύγκρουση συμφερόντων. Το σύστημα αυτό το αναπτύσσουμε μαζί με την Εθνική Υπηρεσία Ακεραιότητας και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι συμπεριλαμβάνουμε όλα τα δεδομένα σε μια διαδικασία δημόσιας σύμβασης. Και έτσι θέλουμε να αποτρέψουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν τη σύγκρουση συμφερόντων και έτσι αποφεύγουμε και τις ε, δημοσιονομικές διορθώσεις εκ των υστέρων. Βέβαια, ε, έχουμε μια μακρά διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απλοποιήσουμε τη διαδικασία, διότι έχουμε πάρα πολλούς ε, φορείς, πολύ λίγους όμως που τελικά αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και αυτό θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να είναι σαφές ε, σε ποιον ανήκουν οι ευθύνες. Ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να μας βοηθήσει πολύ στην ε, περιφερειακή αυτή αναδιάρθρωση και θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους τους ευρωβουλευτές με εμπειρία στον τομέα της αποκέντρωσης να μας βοηθήσουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή που είναι τόσο σημαντική για τη χώρα μας. Όσον αφορά τις μακροοικονομικές προϋποθέσεις, γνωρίζουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι οι προϋποθέσεις αυτές ε, μας επηρεάζουν πάρα πολύ. Για χώρες όπως είναι η Ρουμανία ε, ε, υπάρχει το θέμα Είναι θέμα να μην, να μην ε, τιμωρηθούμε δύο φορές για το ίδιο θέμα. Ε, και έχουμε το θέμα της ε, περιφερειοποίησης. Όσον αφορά την επικάλυψη εργασιών, έχουμε μία διυπουργική επιτροπή η οποία ασχολείται με το θέμα της αποκέντρωσης. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιος θα κάνει τι και Ελπίζω να ε, σταματήσουμε να έχουμε ε, μοιρασμένε αρμοδιότητε στη Ρουμανία, διότι όταν είναι πολύ υπεύθυνοι τελικά κανεί δεν είναι υπεύθυνο. Ε, θα προσπαθήσουμε να υποβάλουμε σε εσά και σε άλλου συναδέρφου σα πληροφορίε σχετικά με όλα τα μέτρα που αναλαμβάνουμε και όλε τι προσπάθειε που καταβάλουμε, διότι ο χρόνο είναι πολύ σύντομο. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που μα δεχτήκατε εδώ και που μα δώσατε την ευκαιρία να σα δείξουμε τι προσπαθούμε να κάνουμε στο πλαίσιο αυτής της πολύ σημαντικής διαδικασίας ε, αποκέντρωσης ε, που πραγματοποιείται στη Ρουμανία. Σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις σας, ε, διότι μου δείχνουν ότι σας ενδιαφέρουν αυτά που πραγματοποιούνται στη Ρουμανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους ε, όλων των ε, συναδέρφων ε, που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και που μοιραστήκατε μαζί μας τα σχέδια σας για να αντιμετωπίσετε όλα τα προβλήματα. Ε, διαπιστώσαμε την ε, αφοσίωσή σας ε, όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις και την, τις προσπάθειές σας για να απορροφηθούν όλοι οι πόροι από τη Ρουμανία. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και θέλουμε να σας πούμε ότι είσαστε ανα πάσα στιγμή ευπρόσδεκτη στην Επιτροπή μας. Καταλαβαίνουμε από την άλλη ότι απομένει να γίνει πάρα πολλή δουλειά. Ευχόμαστε ότι καλύτερο και ελπίζουμε να έχετε επιτυχία στη Ρουμανία με όλες τις προσπάθειές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Dear colleagues, we immediately start. Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μα. Έχουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη το σημείο 14. Πριν όμω περάσουμε σε αυτό, θα ήθελα να σα ανακοινώσω τι αποφάσει που ελήφθησαν χτες από του συντονιστέ. Κατά τη διάρκεια τη συνεδρίας των συντονιστών, σε ό,τι αφορά την ε, κατανομή εκθέσεων, γνωμοδότηση για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για το σχέδιο δράση για την ηλεκτρονική υγεία ε, δόθηκε στο EDF. Η έκθεση ίδια πρωτοβουλίας μάλλον ε, ακολουθήσαμε Όσο είχαμε αποφασίσει το Φεβρουάριο, οι φιλελεύθεροι και γκουε πρότειναν αναθεωρημένη έκθεση της ε, για τη συνεδρίαση των συντονιστών του Απριλίου. Οι συντονιστέ επίση αποφάσισαν ότι η έκθεση της πρωτοβουλία θα ζητηθεί άμεσα όταν η έκθεση του κυρίου Βλάσακ υιοθετηθεί, που ελπίζω ότι θα είναι το Μάιο, και ταυτόχρονα συστήσαμε σε όλους τους συντονιστές και μίλησαν ε, με τους συζητητές ε, των συνεχιζόμενων εκθέσεων να επιταχύνουν το έργο τους προκειμένου να ελευθερωθεί τουλάχιστον ένα σλότ πριν από τον Ιούνιο. Και αυτό σχετίζεται με το εξής η δυνατότητα υιοθέτηση νέας πρότασης για έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας θα είναι το, κατά τη συνάντηση του Ιουνίου. Τότε θα έχουμε την τελευταία ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Μέχρι τις 20 Ιουνίου δηλαδή. Και επίσης συμφωνήσαμε ότι θα ζητήσουμε από τη διάσκεψη των Προέδρων να κατανέμουν στη Ρέτζη μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλία, μάλλον ένα τέτοιο σλότ εκτός ποσόστοσης, προκειμένου να προετοιμαστεί η έκθεση για τη μελλοντική ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και το ρόλο της νέας πολιτικής συνοχής. Και πιθανή συγκήτρια είναι η πρόεδρό σας. Επίσης, συμφωνήσαμε να ζητήσουμε μια εξωτερική μελέτη για το ίδιο θέμα, για τη διακυβέρνηση και την πολιτική συνοχής και θα ζητήσουμε από το Τμήμα Πολιτικής να το φροντίσει. Επίσης, συμφωνήσαμε σε μια ακόμα εκδήλωση σε σχέση με αυτό το θέμα της διακυβέρνησης και της ε, πολιτικής συνοχής. Αν ε, δεν λάβουμε αυτή τη δυνατότητα να έχουμε μία έκθεση εκτός ποσόστοσης ε, θα έχουμε μία προφορική ερώτηση με ψήφισμα για το ίδιο θέμα και θα μπορούσαν να συμμετάσχουν ε, και άλλες ενδιαφερόμενες επιτροπές για να μπορούμε να κάνουμε μια καλή συζήτηση μετά το καλοκαίρι. Σε ό,τι αφορά τώρα τις Open Days, ε, ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα. δεν μπορούμε να έχουμε την τελετή έναρξης που παραδοσιακά έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί φέτο, η εβδομάδα αυτή συμπίπτει ακριβώ με την εβδομάδα που έχουμε την πρόσθετη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Και προσπαθήσαμε τα πάντα, αλλά είναι αδύνατο να, να αλλάξουμε τι ημερομηνίε για οποιαδήποτε από αυτέ τι εκδηλώσει, δηλαδή ούτε για τι Open Days ούτε για την Ολομέλεια. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να ζητήσουμε τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να δώσει άδεια στον πρόεδρο να έρθει στις Βρυξέλλες για την ενεργητήρια τελετή και μπορεί να ζητήσουμε και πρόσθετη άδεια για όλα τα μέλη της Επιτροπής, Ρέτζι, που θα ήθελα να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις στα εργαστήρια. Αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν από τους συντονιστές χθες. Έτσι λοιπόν, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, εγκρίνονται. Τώρα να δώσουμε το λόγο στους Λαμπέρ και Κωνσταντσα για να μας πείτε που βρισκόμαστε σε σχέση με τον τριμερή διάλογο. Ποιος θα ξεκινήσει. Παρακαλώ, Λάμπερτ. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα θέλω να με ακούν όλοι. Και το θέμα είναι σημαντικό, αρκεί να δείτε πόσα είναι τα έγγραφα και πόσο πολύπλοκα. και χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επιτροπή μας συνεχίζει τη στήριξη της δουλειάς αυτής. Πρέπει να σκεφτούμε τον τρόπο εργασίας μας και το χρονοδιάγραμμά μας. Την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια είχαμε το ψήφισμα για το Πολδίπ που περιέχει πολύ σημαντικά σημεία για την ευελιξία, για τις πληρωμές, τις προβλέψεις κλπ. και πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση. Αν περάσει η θέση του Κοινοβουλίου για τα επόμενα 7 χρόνια, τότε πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερα να έχουμε αποτελέσματα, δηλαδή την νομοθετική πρόταση, να το έχουμε κάπου έτοιμο στο μυαλό μας. Μετά θα δούμε συγκεκριμένα πώς θα το κάνουμε. Σε λίγο θα σας πω λεπτομέρειες. Υπάρχει πρώτα το κεφάλαιο CSF και μετά το κεφάλαιο της περιφερειακής ανάπτυξης. Αλλά γενικότερα μας δώσατε την εντολή εδώ στην Επιτροπή να το εξετάσουμε και να πάμε μετά πριν τις θερινές διακοπές να το περάσουμε στην Ολομέλεια. Πρέπει να δούμε αν μπορεί να επιταχυνθεί, αλλά είναι ρητορικό το ερώτημα. Το λέω και για τον εαυτό μου τον ίδιο, αλλά πρέπει να γίνει μία ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση στην Επιτροπή μας για να δούμε τι πετύχαμε και αν δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία παρόλα αυτά μπορεί να υπάρχουν επιμέρους συμφωνίες. Ίσως να καταλήξουμε σε μια ανάγνωση, αλλά αφού είδα τι έβαλε το Συμβούλιο στο Πολδίπ, το αμφισβητώ. Αν θα μπορέσουμε να έχουμε πλήρη συμφωνία πριν το καλοκαίρι δηλαδή. Γιατί δεν θέλουμε αυτήν τη λεγόμενη performance reserve. Αυτά είναι τα δύσκολα και αν θέλουμε να ψηφίσουμε πριν το καλοκαίρι και να συμμετάσχουν όλοι, ίσως και σε δεύτερη ανάγνωση, πρέπει να βιαστούμε. Εντάξει, είναι πολύ δωρικό ερώτημα, αλλά θα το δούμε και αυτό. Πώς θα επιταχύνουμε λοιπόν για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ώστε να έχουμε αποτελέσματα όσο το δυνατόν συντομότερα. Θα πω λοιπόν δύο πράγματα και μετά θα μιλήσει η συνάδελφός μου και συνεισηγήτρια Κωνσταντσα. Το CSF δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Άρα κατά τα 97% ναι. Και αν θυμάστε, το Κοινοβούλιο καθόρισε τη νομική βάση και έπεισε και τους υπόλοιπους εταίρους του. Αυτό ήταν κάτι καινούργιο στον τρόπο εργασίας μας. και αυτό πέρασε ήδη. Στείλαμε, σας στείλαμε όλες αυτές τις συμφωνίες και ε, concrete to this. Και θα μπορούσαν βέβαια να υπάρξουν καλύτεροι ορισμοί για επίπεδα αναχώρα, για συστάσεις για τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης. Έτσι κάνουμε τώρα. Και οι χώρες και η Ένωση. Και ο στόχος του 2020 με τη συνοχή. Και συζητήσαμε πώς θα προσαρμοστούμε αν χρειαστεί περισσότερη ευελιξία. Το Συμβούλιο είπε σε χωριστό έγγραφο και αμέσως βγάλτε μερικά κομμάτια από αυτό το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και βάλτε τα εκεί. Εμείς δεν το δεχτήκαμε αυτό. Μάλιστα είπαμε ότι ίσως αν χρειαστεί να το κάνουμε με κατεξουσιοδότηση πειράξη. Και ελπίζουμε να το δεχτεί και αυτό το Βούλιο σε αυτό το τελευταίο 2% της διαπραγμάτευσης. Δεν δεχτήκαμε λοιπόν την αποδυνάμωση. Γενικά. κάτι παραμένει ακόμη εκρεμές αλλά δεν είναι κυρία θέματα όλα αυτά. Και το πρωί Κωνσταντσα ήδη είπε ότι δεν συζητήθηκαν τα θέματα ή τα διακυβέρνησης. Εγώ χαίρομαι προσωπικά γιατί μπορέσαμε να επιτύχουμε συμφωνία για κάτι καινούριο, για τη Smart Specialization που συνδέει το πρόγραμμα ορίζων με τα νέα κονδύλια συνοχής και επενδύσεων. Τα κράτη είχαν πει ότι δέχονται τομεακές προτάσεις να συνδυαστούν αυτές και να σταλούν ως δέσμοι για την εταιρική συμφωνία. Εμείς είπαμε όχι, δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη άποψη για όλα αυτά και να προταθεί και με πιο ολοκληρωμένο τρόπο και όχι σαν μπάλωμα και κουρελού. Και αυτό ξεπερνάει και αυτά που αρχικά είχε προτείνει η Κομισιόν. Το ίδιο έγινε και για άλλα θέματα λοιπόν. Τώρα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Εδώ το Κοινοβούλιο δεν πρότεινε δικά του καινούργια στοιχεία, αλλά θέλησε απλώς να κρατήσει το Συμβούλιο στο σωστό δρόμο. για να σεβαστεί την εντολή που είχε αναλάβει. Θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι διατυπώσεις βέβαια και υπάρχουν και μερικά άρθρα που ακόμη συζητιούνται. Ιδιαίτερα για ορισμένες έννοιες όπου τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να μιλήσουν καθόλου για ορισμένες και αυτό παλεύουμε ακόμα. Αλλά αυτά σύντομα θα καταλήξουν. Το 98% τελείωσε και γι' αυτόν τον λόγο άρχισα λέγοντας πώς μπορούμε να φέρουμε τα αποτελέσματα αυτά στην ψηφοφορία. Αν το 98% έχει συμφωνηθεί. Τότε τα εκρεμή θέματα, ιδίως από τα δημοσιονομικά, θα μπορούσαμε να τα ψηφίσουμε σε άλλη φάση. Πρώτα τα κυριότερα όπου έχουμε συμφωνήσει. Γιατί έχουμε προτεραιότητες και ξέρει κανείς τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν. Τα άλλα είναι διαχειριστικά. Τα κυριότερα λοιπόν, ιδίως με το πολζίπ τα έχουμε συμφωνήσει και για τα άλλα νομίζω ότι θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Ελπίζω και η Κωνσταντσα να δέχεται αυτά που λέω σήμερα, όπως και τις άλλες φορές, δεν ξέρω όμως. Άσε να, στα πω, να μας τα πει μόνη της. Ναι, φυσικά περιμένω να μου δώσετε το λόγο, ναι φυσικά συμφωνώ με τον Λάμπερ και δεν θέλω να επαναλάβω όσα είπε. Μία γενική παρατήρηση μόνο θέλω να κάνω, προτού προχωρήσω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως ήδη είπα με τον Επίτροπο Χάν και όπως είπε και ο Λαμπέρ τώρα, μερικές φορές φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου ζητάμε να γίνει χρήση της ηλεκτρονικής συνοχής, ε, όχι μόνο να εφαρμοστεί, ε, μερικές φορές αναρωτιόμαστε τι γίνεται κατά τη διάρκεια του τριμερού διαλόγου. Φαίνεται να είναι κάτι μικρό και απλό, αλλά είχαμε σκληρέ διαπραγματεύσει για την εντολή μας και το Κοινοβούλιο είναι ανοιχτό απέναντι σε συμβιβασμούς. Ε, κοιτάμε το περιεχόμενο, προσπαθούμε να δούμε πού μπορούμε να βρούμε ε, συμβιβασμούς ε, με το Συμβούλιο. Όπως είπε ο Λαμπέρ, έχουμε συμβιβασμούς ε, και το λέμε λοιπόν γιατί θέλουμε να προωθήσουμε κάτι και όχι να το χρησιμοποιήσουμε κιόλα. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στην κατάσταση όπου η Προεδρία λέει Εντάξει, αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην εντολή μου, θα πρέπει να επιστρέψω να ρωτήσω τα κράτη-μέλη. Αυτή λοιπόν είναι μια δύσκολη κατάσταση την οποία δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί δημιουργεί τόσες δυσκολίες η διαδικασία αυτή για τα κράτη-μέλη και γιατί δεν μπορούμε να επιταχύνουμε τις διαπραγματεύσεις ε, στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Τη στιγμή που έχουμε ακόμα πέντε θεματικές ομάδες ανοιχτές, την εδαφική ανάπτυξη, την ε, εκ των προτέρων ε, προϋποθετικότητα κλπ, Ξεκινάμε τώρα, συζητάμε την παρακολούθηση και αξιολόγηση. Στη θεματική συγκέντρωση λοιπόν είχαμε ε, τριμερή διάλογο στις 10 Ιανουαρίου και ακόμα περιμένουμε την πρόταση της Προεδρίας. Εντάξει, μπορεί αυτό να είναι κάπως πιο δύσκολο θέμα, αλλά Θέλουμε να προχωρήσουμε από το σημείο 7 στο 4, την πρόθεση της, ε, των βιώσιμων μεταφορών. Δεν είναι δυνατόν εδώ και 8 εβδομάδες να πάρουμε απάντηση από τα κράτη-μέλη. Εάν συνεχιστεί αυτό και τις επόμενες εβδομάδες, δεν θα... Δεν προλάβουμε να τελειώσουμε αυτό το τέλος της χρονιάς ε, τον κανονισμό. Θα πρέπει λοιπόν να το καταστήσει αυτό σαφές το Κοινοβούλιο και μαζί με τη διαπραγματευτική ομάδα ετοιμάζουμε, προετοιμάζουμε πολύ προσεκτικά κάθε τριμερή διάλογο. Γι' αυτό όμως πρέπει εδώ στην Επιτροπή μας και με την διαπραγματευτική ομάδα να συζητήσουμε πώς θέλουμε να προχωρήσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Να φτάσω σε άλλο θέμα όσον αφορά την ε, θεματική συγκέντρωση. Δεν υπάρχει ε, συμφωνία όσον αφορά το 84-3. Πρόκειται για τις ποσοστώσεις ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ε, δεν έχει κλείσει το θέμα αυτό. Το Κοινοβούλιο έχει εντολή, η Επιτροπή έχει υποβάλει ε, πρόταση και το Συμβούλιο έχει εντολή. Ε, απέχουμε πολύ από την εξέβρεση συμβιβασμού. Γι' αυτό ρωτάμε σήμερα την Κομισιόν εάν υπάρχει κάποια δυνατότητα συμβιβασμού. Δεν έχουμε λάβει απάντηση. η κατάσταση είναι ίδια και εδώ. συμφωνήσαμε και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά θέματα να έχουμε 10% κοινή χρηματοδότηση από το ESF και το ERDF. Ε, άρθρο 8, νομίζω ότι αυτή είναι... Ε, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ θετικό για το Κοινοβούλιο. Ε, υπάρχει μια σειρά εγγράφων με τα αποτελέσματα του τριμερού σε διαλόγου. Μπορείτε λοιπόν να το διαβάσετε αυτό προσεκτικά. Και να δείτε τι έχει αποφασιστεί και τι όχι. Όσον αφορά το ESF και την εδαφική ανάπτυξη, ο Λαμπέρτα είπε όλα. ένα θέμα εκκρεμεί. Θέλουμε οδηγό για τους δικαιούχους και ψάχνουμε το κατάλληλο σημείο στον ε, κανονισμό να έχουμε κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι εύκολο για την Προεδρία να υποβάλει πρόταση. Κατόπιν έχουμε το θέμα πλαίσιο απόδοσης 19-20 ε, και παράτημα 2. Το θέμα εδώ δεν είναι η απόδοση αυτή καθ' είναι το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και στο άρθρο 19 παράγραφος 1 Έχουμε πρόταση του Συμβουλίου. Έχουμε το 2019 μια ημερομηνία αναθεώρησης αντί για το 2017 και αυτό είναι ένα τέτοιο παράδειγμα και το δεχτήκαμε αυτό στο πνεύμα συμβιβασμού και ευελιξίας από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι Κατά τα άλλα, γνωρίζετε πόσο σημαντικά είναι τα θέματα των ε, αναθεωρήσεων για μας, της ημερομηνία αναθεώρησης. Είναι συμβασμός όμως. Ε, η απόφαση για το 19.2, καθότι εξαρτάται από συμφωνία πάνω στο άρθρο 44, παρακολούθηση και αξιολόγηση. Συμφωνήσαμε να αλλάξουμε τον τίτλο του άρθρου 20 να λέμε εφαρμογή ε, αντί για ε, κατανομή του πλαισίου απόδοσης και στο άρθρο 20 περιμένουμε συμφωνία, το 18 το έχει διαγράψει το Κοινοβούλιο. Ε, αυτό συνδέεται και με το άρθρο που έχει να κάνει με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα ε, συζητηθεί αργότερα στις διαπραγματεύσεις. Ε, όσον αφορά το άρθρο 20 και το πλαίσιο, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Υπάρχει τελείως διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τις προθεσμίες. Και περιμένουμε πρόταση από την Κομισιόν για να μπορέσουμε να συνενώσουμε τις ε, διάφορες ε, γραμμές και να δούμε πόσο γρήγορα μπορούμε να πετύχουμε συμβιβασμό. Η εντολή του Κοινοβουλίου προβλέπει ότι αρκεί το τρίμηνο για τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία πάνω στο θέμα αυτό αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά το 20 παράγραφος 4 υπάρχει συμφωνία σχετικά με το τι είναι αυτό και τι διορθωτικές πράξεις θα γίνουν. Στο παράρτημα 2 ε, έχουμε τη μέθοδο για το πλαίσιο απόδοσης. Μπορεί να βρούμε ε, τελικά συμβιβασμό σχετικά με τον ε, ορισμό, με τους διάφορους ορισμούς μόνο όμως για τα χρόνια 2018 και 2022, όχι όμως για το 2016. Αυτό συνάδει με τον κανόνα νη συν 3. Ε, που ε, συζητήθηκε στο, στη Σύνοδο Κορυφής αρχές Φεβρουαρίου. Επίσης, Έχουμε ε, το θέμα της εκ των προτέρων προϋποθετικότητας. Ε, εδώ η πιθανότητα να υπάρξει συμβιβασμός με βάση την αρχή ότι η αναλογικότητα θα εφαρμοστεί όσον αφορά την ε, διόρθωση και την αναστολή των πόρων αλλά όχι όμω για τη διόρθωση της ε, εκ των προϋποθετικότητας. Ε, το Συμβούλιο ε, ανέλαβε να υποβάλει σχετική πρόταση και περιμένουμε και την, την οποία περιμένουμε ακόμα στο παράρτημα 5 και όπου έχουμε την θεματική εκ των προτέρων προϋποθετικότητα σε πολλά σημεία το κείμενο πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το παράρτημα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Συχνά έχουμε πιο ήπια διατύπωση από πλευρά του Συμβουλίου ε, αναφέρεται σε αποτελέσματα αντί για ε, και διάφορα άλλα τέτοια. Μπορούμε να το δεχτούμε αυτό ή όχι, αλλά αν μπορεί η Κομισιόν να το δεχτεί, τότε μπορούμε και εμείς στο πνεύμα συμβασμού να ακολουθήσουμε την πρόταση. Εκκρεμούν ακόμα κάποιες ερωτήσεις, όπως στον στόχο 3, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Το Συμβούλιο έχει διαγράψει την αναφορά σε συγκεκριμένου στόχους και πολύ συχνά η διαγραφή των κριτηρίων ε, ή των, ε, αναφορών, των σημείων αναφοράς ε, έχουν χαλαρώσει ή έχουν διαγραφεί. Ε, και, στις, ε, και στη Γενική Εκ των Προτέρων Προποθετικότητα δεν έχουμε βρει ε, συμφωνία πάνω στο θέμα αυτό, καθότι το Συμβούλιο θέλει να διαγράψει σχεδόν το σύνολο του κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένη τη Εκ των Προτέρων Προποθετικότητα όσον αφορά την ισότητα των φύλων, τα ίσα δικαιώματα για αναπήρου κλπ. Και έχουμε πει ότι αυτό για το Κοινοβούλιο σαφώ είναι μια κόκκινη γραμμή την οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να ε, βρούμε συμφωνία, αλλά ε, το Κοινοβούλιο έχει πολύ σαφή θέση στο θέμα αυτό. Συμφωνία πάνω σε κάποιες ε, πτυχέ τη προποθετικότητα για τις δημόσιε συμβάσει, τι κρατικέ ενισχύσεις, το στατιστικό σύστημα κλπ. Μπορούμε να συζητήσουμε αν το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Είμαι πάντα αισιόδοξη, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε συμβιβασμού τις επόμενες μέρες και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε κάποια, ε, κάποιες δέσμες θεμάτων και να ανοίξουμε κάποιες άλλες και να προχωρήσουμε. Αύριο η διαπραγματευτική ομάδα θα πρέπει να συζητήσει τη διαδικασία για τις επόμενες εβδομάδες. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε στις αρχές του Μαΐου να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ε, τα τελικά αποτελέσματα στις περισσότερες δέσμες θεμάτων. Ευχαριστώ η Ελίζα Σέτερ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ε, να αναφερθώ στο οροκλήμα, διότι υπόθηκαν ε, ήδη πολλά. Έχουμε την εξής κατάσταση. Από τη μία μεριά θέλουμε να προχωρήσουμε, διότι έχουμε ευθύνη για το σύνολο της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων αυτών, το είπε ο Λαμπέρ. Από την άλλη μεριά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, διότι επιμένει το Συμβούλιο. Σε όλες τις προτάσεις που υποβάλλει το Κοινοβούλιο λένε όχι. Ακόμα και αν προσπαθήσουμε να πούμε ότι ωραία, συμφωνούμε σε ένα μέρος, υπάρχουν δύο-τρία θέματα όπου έχουμε διαφορετική θέση. Μήπως μπορούμε να βρούμε κοινή συμφωνία, ο ένας να πάρει αυτό, ο άλλος το άλλο. Έχω την εντύπωση ότι σε όλα λένε όχι. Ουσιαστικά ούτε αυτή τη δυνατότητα δεν έχουμε. Το κοινοβούλιο λέει πρέπει να κλείσουν κάποια κεφάλαια, δεν, μπορούμε να δεχτούμε, δεν, μπορείτε να προσπαθήσετε να ε, το δεχτείτε. Ε, αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε συνέχεια. Ε, πράγμα που δυσκολεύει πολύ τη ζωή, την ε, ζωή της ε, διαπραγματευτικής ομάδας. Ε, λέμε ότι ωραία, σχεδόν έχουμε καταφέρει αυτό που θέλαμε, αλλά το Συμβούλιο δεν μετακινείται, οπότε να μετακινηθούμε εδώ. εάν λοιπόν κάποια στιγμή πούμε ότι όχι, δεν θέλουμε να μετακινηθούμε, τότε το Συμβούλιο λέει ότι α, δεν μας ενδιαφέρει. Ε, λέμε ωραία η, η Κομισιόν να υποβάλει συμβαστική πρόταση, το Συμβούλιο διαγράφει όλα τα σημεία που δεν θέλει. Έτσι λοιπόν, ε, οποιαδήποτε προσπάθεια να συμπεριληφθούν και οι δύο θέσει ε, στο έγγραφο μπλοκάρονται από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θέλει μόνο το δικό του κείμενο. Το βασικό επιχείρημα του Συμβουλίου είναι ότι πρέπει να ρωτήσω 27 κράτη-μέλη αν συμφωνούν και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και εμεί έχουμε, δεν ξέρω πόσα μέλη έχει η Επιτροπή μα, ε, η Επιτροπή μα 60 άτομα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει και εμεί να ρωτήσουμε 60 ευρωβουλευτέ, αλλά δεν το λέμε αυτό. Λέμε ότι έχουμε μια εντολή η οποία μας δίνει κάποια ευελιξία, διότι ξέρουμε ποια είναι η πρόθεση του Κοινοβουλίου, αλλά το Συμβούλιο δεν λειτουργεί καθόλου έτσι. Εγώ θα έβρισκα χρήσιμο οι συνάδελφοι να σκεφτούν ε, εάν θα πρέπει να είμαστε πιο σκληροί με κίνδυνο να καθυστερήσουμε να χωρίσουμε τη θέση μας ε, ελπίζοντας να προχωρήσουμε ακόμα και αν ε, δεν φαίνεται η θέση μας στο κείμενο. Πιστεύω ότι πρέπει να το πούμε αυτό, διότι η ομάδα ε, ε, συνειδητοποιεί την ευθύνη της όσον αφορά την εντολή, αλλά από την άλλη ε, καταβάλει και υπεράνθρωπες προσπάθειες. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να έχει ζητήσει κανείς άλλο το λόγο. Όλοι είναι ικανοποιημένοι λοιπόν ή ε, μήπως ε, δεν ακούνε τι λέτε. Παρακαλώ Κωνσταντσα. Μία σύντομη παρατήρηση να προσθέσω. Ομολογώ ότι η Ελίσαμπετ δεν έχει άδικο, αλλά νομίζω ότι δίνει κάπως λάθος εικόνα. Ναι, λέμε ότι προχωράμε πολύ αργά, αν κοιτάξουμε το χρονοδιάγραμμα ε, που έχει υποβάλει στο Κοινοβούλιο το Συμβούλιο, είναι πράγματι απίστε... θα ήταν απίστευτο αν το είχαμε πετύχει. Ε, και πάντως δεν ευθύνεται το Κοινοβούλιο που δεν έχουμε ολοκληρώσει το θέμα. Ο Λάμπερτ ε, λέει και μάλιστα σωστά ότι έχουμε διαπραγματευτεί το 95% των θεμάτων σε πολλούς ε, στα περισσότερα θέματα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διάσταση απόψεων. Λίγα είναι τα σημεία όπου υπάρχουν ε, αυτές τι διαφορετικές θέσεις. Ε, το να πούμε ότι δεν πετυχαίνουμε τίποτα είναι λάθος. Μπορεί γι' αυτό να μην έχει πάρει κανεί το λόγο εδώ στην Επιτροπή, διότι μπορεί να, ε, να έχουμε πλημμυρίσει τους συναδέλφους με την έλλειψη ικανοποίησής μας. Είχα τη χαρά να είμαι και στον διάλογο ΕΦΡΑ. Εκεί ε, συστάμε ώρες για μια παράγραφο χωρίς να καταλήγουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Ε, σίγουρα ε, στα γενικά θέματα προχωράμε πολύ πιο γρήγορα. Βέβαια υπάρχουν πολύ περισσότερα θέματα που πρέπει να συζητηθούν εδώ. τα, οι, οι βασικές πολιτικές θέσεις του Κοινοβουλίου δεν ε, έχουν συστηθεί ακόμα. Ε, τι, να σας πω, να αναφερθώ στην μακροοικονομική ε, ε, προϋποθετικότητα. Είναι πολύ αυστηρή η εντολή μας και πώς θα καταλήξουμε σε συμβιβασμό εάν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με πιο, σε πιο ασήμαντα θέματα. Αυτό με ανησυχεί, αλλά ίσως θα πρέπει να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με τέτοιο τρόπο ώστε στο τέλος να έχουμε κάποια θέματα, 2, 4, 6, 8, όπου να μην υπάρχει συμφωνία και τότε να πούμε ωραία τι θα κάνουμε τώρα. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε ή θέλουμε να συνεχίσουμε μέχρι, μέχρι την ημέρα του Αγίου ποτέ. Να δούμε τι θα έχουμε τελικά στο επτάπητο και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, Γιώργη. Συνάδελφοι. Από αυτά που άκουσα ίσως ε, είναι ακριβώς αυτή η τακτική ε, του Συμβουλίου να κολλάει σε ε, ασήμαντα θέματα, να αφήνει το χρόνο να περνάει ώστε όταν φτάσουμε στα σημαντικά θέματα και η Κωνσταντς ανέφερε κάποια από τα θέματα αυτά, να λέει ότι α, δεν έχουμε χρόνο, ε, θα πρέπει πολύ γρήγορα να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Ίσως ε, να αντιστρέψουμε το θέμα και να πούμε ωραία, ας αφήσουμε ε, κατά μέρο τα μικρά θέματα και να κοιτάξουμε τα μεγάλα συμπλέγματα προβλημάτων και να πούμε ωραία ποια είναι η θέση σας για αυτά. Υπάρχει ήδη θέση του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά, διότι αλλιώς, και το ακούμε αυτό και από άλλους ε, γύρους διαπραγματεύσεων, ε, ότι κολλάνε οι συζητήσεις στα ασήμαντα θέματα και τελικά ε, χρησιμοποιεί το Συμβούλιο την πίεση του χρόνου στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε λοιπόν να ξέρουν ε, πώς θα είναι τα πράγματα ε, μετά το 2013. Ε, τα κράτη-μέλη θέλουν να ξέρουν πώς θα διαμορφώσουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Ε, Φοβάμαι λοιπόν ότι δεν περιμένουμε καν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και ότι έτσι τελικά μας μας παραμερίζουν. Ε, δεν νομίζω ότι θα ήθελα να... Ε, νομίζω ότι πρέπει να αντιστρέψουμε το όλο θέμα. Ο Λάμπερ. Ναι, ναι, κουμπί. Εδώ βλέπω το σχεδιασμό του τριμερούς διαλόγου και έχασα το μέτρημα και ζήτησα από τη γραμματεία να μου πει αν έχουμε αύριο τη συζήτηση παριθμών 18 ή 19, αλλά αν το ολοκληρώσω αυτό έχουμε 40. Δηλαδή, πολλά κάνουμε, αλλά που είναι η αποτελεσματικότητα. Επίσης, ίσως ε, να ζητήσουμε από τον πρόεδρο του Μεριστιολόγου να έρθει κάποια στιγμή και να πει στο Συμβούλιο και στους υπουργού ότι θέλουμε να είμαστε έτοιμοι το συντομότερο δυνατόν με ένα καλό αποτέλεσμα. Και αυτό σημαίνει με τη δυνατότητα επιτυχίας. Στο κοινοβούλιο αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να έχουμε μια πρώτη κατάληξη τον Ιούλιο. Δεν είναι τρελό αυτό. Σε ένα χρόνο πρέπει κάποιος να παρουσιάσει αποτέλεσμα ή αλλιώς ε, είναι ανίκανο να κάνει κάτι. Και αν ε, δούμε τη στιγμή στην οποία βρισκόμαστε τώρα, ίσως ε, θα πρέπει να θέσουμε και ένα όριο, να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, όσο είπε ο συνάδελφο ισχύουν, πάντοτε υπάρχουν άρθρα, ολοκληρώνονται, αλλά πάντοτε κάτι ανακύπτει. Μπορεί να υπάρχουν κάποια άλλα που μπορεί να αναφέρει ο καθένας. Ε, να έχουμε 5-6 σημεία το πολύ που θα πάνε στο επόμενο στάδιο Τη δεύτερη ανάγνωσης. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος να πράξουμε και ίσως θα πρέπει να το πούμε και σύντομα στην Προεδρία ότι αυτά είναι τα δικά μας σημεία και αυτές είναι και οι κοκκινέ γραμμές. Έτσι ώστε να καταλάβουν ότι αν εξοδεψουμε πανω πάνω 5-6-7 ημέρες επί των λεπτομεριών, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό στους συναδέλφους, που μπορεί να κινούνται ταχύτερα σε άλλους τομείς. Έτσι λοιπόν, ο καθένας ακολουθεί το δικό του δρόμο, αλλά πρέπει να επιταχύνουμε. Και ίσως ε, θα έπρεπε να σημειώνουμε μία πρόοδο σύντομα. I, I want... Αναρωτιέμαι μήπως η Κομισιόν θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Ναι, ευχαριστώ. Θέλω να κάνω κάποιες ε, σύντομες παρατηρήσεις. Ε, το πρώτο από την σκοπιά της Κομισιόν μας ε, συμφέρει και εμάς να συμφωνηθεί το συντομότερο δυνατό αυτό το πακέτο γιατί θέλουμε να τρέχουν τα προγράμματα σε καιρό κρίσης. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να συνειδητοποιούν τους ενδυνάμει κινδύνους ε, του να κολλήσουμε σε μια δύσκολη διαδικασία. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό και το Συμβούλιο να συνειδητοποιήσει όλους τους κινδύνους. Επίσης, ε, θα ήθελα να επανέλθω σε κάτι που είπε η κυρία Κρέλαν, είναι μισογεμάτο δύο το ποτήρι. Νομίζω ότι ορισμένα από τα δύσκολα ζητήματα έχουν ε, ήδη αντιμετωπιστεί και από τη σκοπιά της Κομισιόν. Όταν βλέπουμε τον προγραμματισμό, τον κώδικα διδοεκλογίας και το ΣΥΣΕΦ, αυτά φαίνονται ε, πάρα πολύ δύσκολα και το γεγονός ότι σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί όλα, με μια δύο λεπτομέρειε απλώ να παραμένουν, είναι κάτι πολύ θετικό. Αυτά είναι τα κυρία στοιχεία που είναι απαραίτητα για να ξεκινήσει ο προγραμματισμός στα κρατημέλη και αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα ε, για την ε, ορμή που μπορεί να δοθεί στην όλη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να υπάρχει προθυμία συμβασμού και από τις δύο πλευρές και από τη σκοπιά της Κομισιόν. Νομίζω ότι έχουμε δει βούληση συμβιβασμού και εμείς έχουμε παρουσιάσει συμβιβαστικά κείμενα και ελπίζουμε τις επόμενες εβδομάδες ότι και το Συμβούλιο θα στείλει ένα τέτοιο μήνυμα γιατί αν δεν δούμε αυτό το μήνυμα σύντομα, τι επόμενε εβδομάδε από το Συμβούλιο, θα βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια. Καταλαβαίνω ότι η λογική των διαπραγματεύσεων είναι σαφής. Θέλουμε να αφήσουμε τα δύσκολα κατά μέρος προς το παρόν γιατί αφού δεν δεχόμαστε τη θέση του Συμβουλίου και το Συμβούλιο δεν δέχεται τη δική μας, πρέπει να αρχίσουμε έτσι. Δεν είναι και πάρα πολλά τα αμφιλεγόμενα. Και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτά και εκτός της δομής του τριμερούς διαλόγου. Να καταλάβει το Συμβούλιο ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα θέματα αυτά όπως είπε και ο Λαμπέρ και ελπίζω και οι, άλλες και οι διάφορες πολιτικές ομάδες να καταλάβουν ποιοι θα είναι οι καλύτεροι δυνατοί συμβιβασμοί γιατί δεν νομίζω ότι δίνουμε την εντύπωση ότι απλώς τα κάνουμε για το Θεαθήνε. Θέλουμε πράγματι να υπάρξει μια ρεαλιστική εφαρμόσιμη πολιτική, όχι υπερβολικά πολύπλοκη. Και εγώ ως προεδρεύουσα του τριμερούς αυτού διαλόγου τους δείχνω πάντοτε ότι θέλουμε να βρεθεί μια πραγματική λύση, ότι δεν το κάνουμε μόνο από πολιτική αντίθεση και διάθεση αντιπαράθεσης. υπάρχουν θέματα όπου πιστεύουμε απλώς ότι η πρότασή μας είναι πιο σωστή και καλύτερη. Δεν θα το αποφασίσουμε βέβαια σήμερα, αλλά πρέπει να έχουμε μια, για να το πω έτσι, σύνοψη της θέσης μας και η Κομισιόν δείχνει καταρχάς να συμφωνεί όχι σε επίσημο τριμερή διάλογο αλλά σε συνεννοήσεις όπου πρέπει να εξηγήσουμε γιατί δεν μετακινούμαστε από αυτές τις θέσεις. Και ίσως έτσι και το Συμβούλιο να καταλήξει να είναι τελικά πιο ανοιχτό. Ξέρω και πώς έχουν γίνει οι άλλοι τριμερείς διάλογοι. Ε, Ξέρουμε ότι το Περιφερειακό Ταμείο είναι πολύ δύσκολης λειτουργίας και πρέπει να προσέχουμε την κάθε λέξη. πολλές φορές προσθέσαμε λεπτομέρειες που είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί. Γιατί ή θα παραμείνει κανείς στο γενικότερο πλαίσιο ή άμα μπει στις λεπτομέρειες πρέπει να τις βάλει όλες. Τώρα όμως και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο απομακρύνθηκαν από την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Και χρειάστηκε να συζητηθούν και παρεμφερεί θέματα όπως το αν οι μεταφορές θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον κλπ. Αλλά δεν χρειάζεται νομίζω να ανησυχούμε για τις λεπτομέρειες. Μπορούμε να τα διευθετήσουμε. Είναι θέμα χρόνου, αρκετού χρόνου. Η πραγματική πρόκληση είναι ε, τα θέματα στα οποία εξ αρχής διαφωνούμε ως θέμα αρχής. Πρέπει λοιπόν να συνεννοηθούμε πράγματι με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για να δούμε σε ποια θέματα δεν θα μετακινηθούμε για την κατανομή των κοντιλίων του Κοινωνικού Ταμείου και τα ακριβή κριτήρια που θέλουμε να εφαρμοστούν. Ελπίζω λοιπόν και για τα δύσκολα να γίνουν τέτοιες συνεννοήσεις άτυπου τριμερούς διαλόγου. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι το Συμβούλιο είπε ότι από τα μέσα Μαρτίου θα γίνει η μεταφορά του διαπραγματευτικού κοιτίου και ότι με συναπόφαση μάλιστα θα γίνει αυτή η μεταφορά και δεν την πήραμε ακόμα, δεν την λάβαμε. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν γνωρίζει τίποτα για την τύχη του. Αυτό είναι το ανησυχητικό, γιατί υπάρχουν εκεί σημαντικά θέματα που μπορεί να διαφωνήσουμε. Η performance reserve και το 7% που μπήκε εκεί των πληρωμών του Περιφερειακού Ταμείου μετά το 20 είπε η Κομισιόν ότι το νήσιν 3 σημαίνει 40% των πληρωμών μετά το 20. Αυτά είναι βασικά θέματα ως προς τις επιπτώσεις που θα έχουν στον προϋπολογισμό αν αποφασίσουμε να τα αλλάξουμε, να βάλουμε το απόθεμα στο, από το 7 στο 5% ή από το 5 μετά στο 0%, αυτά έχουν μεγάλες σοβαρές επιπτώσεις στο επίπεδο των πληρωμών για το 14 με 20. Και αυτό δεν είναι παρά ένα παράδειγμα. πολύ δύσκολα θέματα όλα αυτά γιατί δεν έχουμε πάντα μόνο την εντολή της Περιφερειακής Επιτροπής αλλά και τα αποτελέσματα ψηφοφοριών της Ολομέλειας. Και αυτό ισχύει και για την μακροοικονομική, ε, για το μακροοικονομικό σχεδιασμό και τους όρους που του έχουμε βάλει και το τι θα, πώς θα γίνει η κατανομή μεταξύ των ταμείων. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όταν θα, ζητήσουμε, θα αναζητήσουμε τους συμβιβασμούς. Πάντως δεν είναι τα πράγματα τόσο άσκημα όσο τα λέμε μερικές φορές. Νομίζω ότι κινούμαστε αρκετά γρήγορα. Και αυτά που είπε ο Πίτερ είναι παρήγορα. Ελπίζω λοιπόν να τα καταφέρουμε παρά τους αρνητικούς μέχρι τώρα δείκτες. Έχει κανεί σχόλια επ' αυτόν, αν όχι, να περάσουμε στο επόμενο που είναι το Περιφερειακό Ταμείο. Γιάνν Όλμπριχτ όμως απουσιάζει. Αλλά μου έδωσε ένα σημείωμα να σας το διαβάσω. Να σας πω ότι αυτός ο κανονισμός είναι ακριβή πάρα πολύ δύσκολος επειδή έχει λεπτομερή φύση και προσπαθεί να εξεύρει την, το να εξεύρουμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ όλων αυτών λεπτομεριών είναι πολύ δύσκολο. Όμως νομίζω ότι κάναμε ουσιαστική πρόοδο επί του πεδίου εφαρμογή για τα θέματα της ε, ενίσχυσης, τα περισσότερα έχουν συμφωνηθεί. Υπάρχει όμως ένα πολύ δύσκολο θέμα που δεν έχει κλείσει ακόμη και είναι η πρόσβαση των μεγάλων επιχειρήσεων στην ενίσχυση, στην υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή. Είμαστε κοντά στο συμβασμό, δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμη. Τα περισσότερα θέματα βέβαια έχουν συμφωνηθεί σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες επενδύσεων. Ακριβώς εδώ ήμασταν πάρα πολύ δημιουργικοί και εμείς και το Συμβούλιο απομακρυνθήκαμε από την πρόταση της Κομισιόν και εδώ ουσιαστικά αγωνιζόμαστε και προσπαθεί ο ένας να πείσει τον άλλον για μικρά θέματα. Και εδώ έχουμε ένα μεγάλο κατάλογο ανοιχτών ζητημάτων. Κατόπιν για την αστική διάσταση, Urban Dimension, είμαστε πολύ κοντά στο συμβιβασμό και πριν την τελευταία συνάντηση χθε φαινόταν κάτι αδύνατο, δηλαδή η ανάθεση στις ε, ε, αρχές, ε, στις δημοτικές αρχές, έχουμε συμφωνήσει επί όλων των στοιχείων και πιστεύω ότι με νέα πρόταση διατύπωσης της Κομισιόν την επόμενη φορά θα καταλήξουμε στη συμφωνία. Επίσης είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία για την πλατφόρμα για την αστική πλατφόρμα η Προεδρία θα ελέγξει με το Συμβούλιο αν θα μπορούσε να δεκτεί το όρο networking αντί για πλατφόρμα. Είμαστε πολύ κοντά στην τελική απόφαση, γιατί επί της ουσίας έχουμε συμφωνήσει, δηλαδή επί του άρθρου, έχουμε κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με την ονομασία. Έχουμε σχεδιάσει τον επόμενο τριμερή διάλογο στα τέλη Απριλίου και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια δύσκολα θέματα. Πάντως πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στην κρίσιμη μάζα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σχόλια. Παρακαλώ, Λάμπερτ. Ξέρω ότι δεν είναι στην εντολή μας το είναι ότι η υποδομή για το αέριο μπορεί να επιδεχθεί χρηματοδότηση. Άκουσα ότι το Συμβούλιο έχει θεκτική προσέγγιση απέναντι σε αυτό και η Κομισιόν και ίσως ε, θα πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό το σημείο, αποκλείεται στην εντολή, αλλά μπορεί να είναι σημαντικό για ορισμένες χώρες και ίσως ε, και πολιτικά πρέπει να είμαστε ειλικρινεί ε, μεταξύ μας για το αν θα επιμείνουμε σε αυτό ή αν θα προχωρήσουμε. Και πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή και αυτό. Πρόεδρο, εδώ λοιπόν το Συμβούλιο και η Κομισιόν είναι ενωμένοι, ενώ το Κοινοβούλιο είναι από την άλλη όχθη. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Βρήκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τους φιλελευθέρους, εγώ θέλω να επιμείνω σε δύο σημεία. Καταρχήν, το είπε και ο Πρόεδρός μας, ε, η Πρόεδρός εδώ εμπλέκονται και μεγάλε επιχειρήσει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μα ομάδα να μπορούν να υποφεληθούν από αυτές τις ενισχύσει μεγάλε μεγάλες επιχειρήσεις. Όμως, με σαφήνεια λέγεται στην ελληνική καταρχήν μικρέ και μεσές επιχειρήσει. Ε, μα θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη διατύπωση και στο τελικό κείμενο του κανονισμού. Είναι ζήτημα σημαντικότατο. Κάτι ακόμα, σε σχέση με όσο είπε ο Λάμπερτ, για το αέριο ή τις ενισχύσεις ε, για τις ενεργειακές ε, πηγές από ορυκτά καύσιμα. Αναφέρθηκε και το αέριο συγκεκριμένα. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε όμως ε, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι στην ενέργεια από ορυκτές πηγές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της εντολής. Μετά από πολλές συζητήσεις εδώ στο Κοινοβούλιο, εκπονήσαμε μία εντολή, ε, την οποία όμως θα πρέπει να χειριστούμε πολύ προσεκτικά. Δυσάρεστο βρίσκω ότι πολύ γρήγορα εγκαταλείπουμε θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην εντολή μας, ε, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να ανακτήσουμε. Βρίσκω λοιπόν ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Και αναφέρθηκε επανειλημμένα ότι στις διαπραγματεύσεις δίνουμε και κάτι δίνουμε, κάτι παίρνουμε, αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι υπάρχουν κάποια θέματα ε, τα οποία χειριζόμαστε με κάποιον ε, τρόπο ε, που κάποιες πολιτικές ομάδες φαίνεται να βρίσκουν σωστό. Ένα παράδειγμα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ότι θα πρέπει να αποτελέσει κόκκινη γραμμή στις διαπραγματεύσεις, αλλά στις διαπραγματεύσεις βλέπω ότι και εντός της ε, διαπραγματευτική ομάδας υπάρχουν διαφορετικές θέσεις ε, και δεν υπάρχει ακόμα, δεν υπάρχει πάντα συνεννόηση εντός της ομάδας. Αυτό το λέω πολύ προσεκτικά, αλλά είναι κάτι που μας δυσαρεστεί. Επίσης, ε, δεν θέλουμε νέε δομέ. συμφωνούμε όσον αφορά αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τηρήσουμε τη γραμμή αυτή. Θέλουμε δικτύωση, δεν θέλουμε όμως να δημιουργήσουμε νέους φορείς. Θέλουμε να προωθήσουμε τη δικτύωση. Εμείς ως πολιτική ομάδα ήμασταν κατά του συνολικού αυτού θέματος, ε, αλλά ε, μιλάμε για δικτύωση. Να μην έχουμε δημιουργία νέων φορέων. Ξέρετε ότι και η Επιτροπή των Περιφερειών έχει ε, μιλήσει κατά του θέματος αυτού. Σημαντικό είναι οι ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βρίσκω ε, πολύ άσχημο το να μπουν τα καύσιμα από την πίσω πόρτα. Έχουμε συζητήσει ότι πρέπει να έχουν προτεραιότητα οι βιώσιμες πηγές ενέργειας. οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια θα πρέπει να αποστασιοποιηθούμε από το θέμα αυτό, αλλά η διαπραγματευτική ομάδα χρειάζεται σαφή θέση. Πρέπει και εμείς δηλαδή να συνοηθούμε μεταξύ μας. Ε, δεν βλέπω κανένα λόγο να απομακρυνθούμε από αυτά που λέει η εντολή, διότι ε, σχετίζεται με όλα τα θέματα αυτά. Όπως και το θέμα τι θα κάνουμε με τα αεροδρόμια. Είπαμε, ωραία, θα υποστηρίξουμε συγκεκριμένα μέτρα για το περιβάλλον, αλλά διαπιστώνουμε ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να διαπιστώσουμε τι μέτρα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Και για παράδειγμα, αρκεί να, ε, ε, ο όρος air ή πρέπει να μιλάμε για airport, για αεροδρόμιο. αναφέρθηκαν τα θέματα αυτά, αλλά μάλλον ε, δεν έχουμε μείνει σε αυτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπαράτσου. Ε, Ευχαριστώ. Είναι πολύ πιθανό ότι το θέμα που πρόκειται να θέσω είναι πολύ συγκεκριμένο για να συζητηθεί τώρα καθώς λείπει ο εισηγητής όμως είναι ένα σημαντικό ζήτημα και θεωρώ ότι πρέπει να το θέσω ζητώ συγγνώμη αν είναι κατάλληλη χρονική στιγμή γιατί είμαι και καινούργια σε αυτή την επιτροπή έτσι λοιπόν ε, πρέπει να δω και πώς λειτουργεί η ίδια η επιτροπή και ποιο είναι και το περιεχόμενο θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 75 της εντολής για μένα θα ήταν σημαντικό να καταλάβω αν στους διαλόγου. διαλόγους συζητήθηκε μάλλον η τροπολογία 75 για το άρθρο 4 η ομιλήτρια, δηλαδή η αναγνώριση να μπορούν οι ε, περιοχές να επαφελούνται από τη θεματική συγκέντρωση όταν μιλάμε για λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές ή για νησιωτικές περιοχές. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν ιδιαίτερες τοπικές και δαφικές απαιτήσει και συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, να δίνονται περισσότερα κονδύλες σε αυτές τις περιοχές. Έχει αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα στον τριμερή διάλογο και υπάρχουν κάποια κοινοί τόποι περισσότερο παρά διαφωνίε ιδέες. Δηλαδή ε, θα ήθελα να δω σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε για την έγκριση αυτής της τροπολογίας. Κωνσταντς. Ε, ε, ναι. Συμμετέχω στο τριμερή διάλογο για το Περιφερειακό Ταμείο. Πρέπει να πω ότι έχω τελείως διαφορετική θέση από την Κορνέλια. Βρίσκω ότι η, ε, ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται απολύτως σύμφωνα με την εντολή του Κοινοβουλίου. Ε, μένουμε λοιπόν στην εντολή μας και δεν μπορούμε να ε, καταλήξουμε σε συμβασμό εάν δεν μετακινηθεί στις θέσεις του το Συμβούλιο. Όσον αφορά την πρόσβαση μεγάλων επιχειρήσεων στα, στις ενισχύσεις. Είχαμε πολύ έντονη συζήτηση ε, στην ε, Επιτροπή μας. Ε, είναι θέμα που σχετίζεται και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά στην εντολή μας έχουμε πει ότι είναι απαραίτητο και μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε τέτοια ταμεία και ακριβώς αυτό αποτελεί το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων στον τριμερή διάλογο. Αντιθέτως ε, βρίσκω δύσκολο ε, να βάζουμε στην εντολή θέματα τα οποία δεν ε, απλοποιούν τις διαπραγματεύσεις. Ε, δηλαδή όταν η διαπραγματευτική ομάδα πιστεύει ότι μπορεί να εκπληρώσει άλλη μια ε, επιθυμία των πολιτικών ομάδων. Θέλω να ε, υποστηρίξω λοιπόν την καθοδήγηση του Γιάννε που τηρεί πολύ πιστά την εντολή. Πιστεύω ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα, καθώς λείπει και ο εισηγητής, αλλά αν κατάλαβα καλά τα σχόλια της κυρίας Μπαράτσου, ό,τι φορά το άρθρο 4, Είχαμε μόνο μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το άρθρο 4, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, στου επόμενου τριμερεί διαλόγου θα γίνει δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν, έχετε κάποιε ανησυχίε να μιλήσετε στον κύριο Όλμπριχτ πριν από εκείνη την συνεδρίαση. Θα ήταν χρήσιμο κάτι τέτοιο. Τώρα για τα θέματα που έχουν να κάνουν ε, με τα μέτρα φιλικά προς το περιβάλλον. Ε, δεν θυμάμαι ακριβώς ε, τι λένε οι οδηγίε, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν σαφείς ορισμοί για το τι είναι φιλικό προς το περιβάλλον ή όχι. Και φυσικά όταν μιλάμε για μικρά προϊόντα δεν θα γίνει τέτοιου είδους αξιολόγηση, αλλά είμαι σίγουρη ότι η Κομισιόν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τα κράτη-μέλη θα ξεκαθαρίσει τι είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τι δεν είναι. Γιατί δεν ε, εμπλέκεται μόνο η ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ ΡΙΤΖΙΟ σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά και άλλες ε, γενικές διευθύνσεις θέτουν ε, σε εφαρμογή επιχειρησιακά προγράμματα. Και Αυτές γνωρίζουν τους ακριβείς ορισμούς. Έτσι λοιπόν, ακόμη και τον ορισμό του ότι είναι φιλικό προς το περιβάλλον δεν ε, θα μπει στον κρισμό. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει ένα σύνολο κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει μια σειρά ορισμών που θα εφαρμοστούν για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, γιατί συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε η Κωνσταντσα να θυμάστε όταν ε, συζητήσαμε το παιδί εφαρμογή ε, στο ΕΤΜΑ είχαμε αυτή την παραγωγική επένδυση, είπαμε μόνο για τι μικρέ και μεσέ επιχειρήσει. Και κατόπιν κάναμε μία μικρή παρέκκληση για τι μεγάλε επιχειρήσει ε, μόνο για πολύ συγκεκριμένε προτεραιότητε, τρει στον αριθμό. δηλαδή το ICT, χαμηλά σε κουβές άνθρακας και γενοτομία. Ακόμη και για το ICT μόνο, όταν ε, υπάρχει το αποτέλεσμα της συνεργασίας ε, μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΜΕ. Γιατί είναι σημαντικό για πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στις ε, διεθνείς αλυσίδες προμήθειας. Και αυτό είναι δύσκολο αν δεν συνεργαστούν με μεγάλες επιχειρήσεις που εργάζονται επί διάφορων θεμάτων. Αυτό είναι ζωτική σημασία. Έτσι λοιπόν, το να στερήσουμε απολύτω το δικαίωμα από τις μεγάλες επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, δεν θα εξυπηρετήσει τελικά την οικονομία. Αυτό αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό το άνοιγμα είναι ζωτικό. Και ήταν και η θέση των κρατών μελών αλλά και της Κομισιόν. Η οποία συμφώνησε με αυτή την προσέγγιση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ακόμα. Για τα υπόλοιπα σχόλια θα περιμένουμε τον εισηγητή, αν συμφωνείτε. Αλλά θα ήθελα, θα σας θαρρύνω να συζητήσετε με τον εισηγητή, αν έχετε περαιτέρω αμφιβολίες, αλλά εγώ την έχω την ίδια τύπωση με την Κωνσταντσα, ότι πρέπει να μείνουμε στην εντολή και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο. Εμεί σεβόμαστε στην εντολή, ενώ το Συμβούλιο μένει στη διατύπωση. Λοιπόν, να κλείσουμε για το έτπα. Και νομίζω η Ρίκα είναι η επόμενη, έτσι. Όχι, ο Βίκτορ. Σας ευχαριστώ, Ντανούτα. Αγαπητοί συνάδελφοι, με τον κανονισμό του Ταμείου συνεχίσει είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, θα έλεγα. Ομαλά, ομαλή ήταν η διαδικασία και μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένο. Να σας αναφέρω ποια είναι η κατάσταση. Μετά την 27 που είχαμε το δεύτερο τριμερή διάλογο, κατορθώσαμε να συζητήσουμε τα ακόλουθα σημεία. Του δείκτε ε, υπαριθμών 2, τι μεταβατικές διατάξει άρθρο 5, το 6, κατάργηση του κανονισμού, το 3 και το 4, θέσει ισχύου του κανονισμού και αναθεώρηση. Επιπρόσθετα, είδαμε κάποιε διατάξει που είχαν αφαιθεί ανοιχτέ από την προηγούμενη συνεδρίαση. Τώρα, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρακτικά ολοκληρώσαμε όλα τα άρθρα του κανονισμού μας στην επόμενη συνάντηση θα επανέλθουμε σε κάποια ζητήματα τα οποία έπρεπε να ολοκληρωθούν και υπήρχαν σοβαροί λόγοι να υπάρχουν σοβαροί λόγοι να θεωρούμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Να πω καταρχήν ότι η διαπραγματευτική ομάδα είναι πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα γιατί ακόμη και αν κάποια θέματα κρεμούν κατορθώσαμε να συμφωνήσουμε σε αρκετά σημαντικά ζητήματα, παραδείγματος χάρη ένα κύριο θέμα ήταν η επιλεξιμότητα της ε, τηλεθέρμανσης και της συμπεραγωγής ε, ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, η διαπραγματευτική ομάδα συμφωνούσε με τον συγητή και το θέσαμε αυτό στις προτεραιότητες επένδυσης και κατορθώσαμε να καταλήξουμε στη συμφωνία με της διατύπωσης που εγγραμμίζεται πλήρως με τις υφιστάμενες διατάξεις στο ΕΤΠΑ μετά τον τριμή διάλογο. Μπορώ να πω ότι η ευθυγράμμιση μεταξύ του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ είναι κάτι που προσπαθούμε να επιδιώξουμε και είναι ένας γενικός κανόνας τώρα. Και η συνεισφορά μας είναι και η συνεισφορά μας για την απλούστευση και για να είναι σαφέστεροι δύο κανονισμοί σε σχέση με τη σειρά των άρθρων τώρα. Οι διαπραγματεύσει ήταν οι εξή. Επιμείναμε στο άρθρο 2, πεδίο εφαρμογή τη στήριξη, παράγραφο για την υποστήριξη που δίνεται από το Ταμείο Συνοχή, ώστε είναι μέσω συνδέοντα την Ευρώπη. Αν μεταβιβαστούν αυτά τα χρήματα, Πιστεύουμε ότι αν πρόκειται να μεταφερθούν αυτά τα χρήματα, είναι προφανέ ότι αυτό θα πρέπει και να αναφέρεται στον κανονισμό του Περιταμείου συνοχή. Επίση, συμφωνήσαμε και η Κομισιόν συμφωνήσε μαζί μα, ότι αν αυτή η διάταξη ευθυγραμμιστεί με το, ε, ότι θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί ε, με τους κανονισμούς για το Connecting Europe Facility. Τώρα, λάβαμε το τελικό εντάξει της Προεδρίας ότι αφορά την επιλεξιμότητα για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για όλες τις επιχειρήσεις, αλλά πρωτίστως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης κατορθώσαμε να συμφωνήσουμε στο να έχουμε ε, την επένδυση για τη συμπαραγωγή ε, θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας και θα είναι επιλέξιμη και η τηλεθέρμανση. Έχουμε μία ε, τροποποίηση για το τομέα του ύδατος έτσι ώστε να διευρυνθούν τέτοιε επενδύσεις και τελικά συμφωνήσαμε επί του κειμένου που λέει ότι το Ταμείο Συνοχής θα υποστηρίξει τις επενδύσεις για, που θα σέβονται τουλάχιστον τις απαιτήσει ε, του Ευρωπαϊκού του περιβαλλοντικού και εκτιμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το Ταμείο Συνοχής θα υποστηρίζει και επενδύσεις που πηγαίνουν παρατέρα στον τομέα αυτό. Αυτό που εκκρεμεί είναι η τελική συμφωνία για το άρθρο 3, για το θέμα των επενδύσεων, για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Γιατί η εντολή μας ζήτησε να, να είναι βασισμένο στο οικοσύστημα. Η Προεδρία δεν φαίνεται να είναι έτοιμη να δεχτεί κάτι τέτοιο και οι επενδύσεις για την ανθεκτικότητα στις καταστροφές θα πρέπει να είναι βιώσιμες. Επίσης, η Προεδρία είπε όχι στη διαπραγματευτική ομάδα και εμείς πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε την επόμενη φορά. Σε ό,τι αφορά τώρα την τροπολογία μας ε, για την ε, ολοκλήρωση και τη συμπληρωματικότητα των επενδύσεων που υποστηρίζεται από διάφορα ταμεία για το τομέα TNT, ε, κάναμε μία πρόταση που ουσιαστικά στην πράξη στο περιεχόμενο συμφωνήθηκε από την Κομισιόν και το Συμβούλιο Τώρα, εγώ είμαι αισιόδοξο ότι θα εγκριθεί η πρόταση κατά τον επόμενο τριμερή διάλογο. Το πρόβλημα που αναμένεται να ανακύψει αφορά τους κοινού δείκτες. Χτες είχαμε μια άτυπη συνάντηση με όλους τους εισηγητές για τους κοινού δείκτες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ίσως η Κωνστάνση και ο Λάμπερτ ε, σας ενημέρωσαν ε, για τις λεπτομέρειες, όμως το πιο σημαντικό είναι η ετοιμότητα του Κοινοβουλίου να συνεργαστεί με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο για μια ευέλικτη λύση που πιθανότατα θα είναι μια καταξουσιοδότηση πράξη για τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στους κοινούς δείκτες, αλλά να συμπεριλάβουμε και στον κανονισμό μας διατάξεις που εκφράζουν τις κυρίες προτεραιότητες για τους κοινού δείκτες ως προς ε, τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχουν. Αυτό είναι τα πιο σημαντικά σημεία. Και τέλος, και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη τη διαπραγματευτική ομάδα για την ε, ενωμένη στάση που επέδειξε στον επέρασπιστή την εντολή μας. Και ελπίζω ότι μετά το τελευταίο τριμερή διάλογο που θα είναι πιθανότητα και ο τελευταίος, να επανέλθω εδώ στην Επιτροπή και να σας πω ότι εκπληρώθηκε η αποστολή μας και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ευχαριστήσα τον πρόεδρο, μόνο ότι είναι διαπραγματευτική ομάδα, αλλά εντάξει. Ο Βίκτορ βέβαια είναι πολύ αισιόδοξο, αλλά η μακροοικονομική προϋποθετικότητα θα εξαρτηθεί από το σύνολο της προόδου. Και... και ελπίζουμε να πετύχουμε συμφωνία όσον αφορά της κατεξοδότηση πράξης ε, και την ε, ανάθεση αρμοδιοτήτων. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλος να σχολιάσει η Κομισιόν θέλει να σχολιάσει. Δεν ε, ρώτησα αν έχετε παρατηρήσεις και για το Περιφερειακό Ταμείο, εάν όχι. Κορνέλια, παρακαλώ. Ναι, πολύ σύντομα. Ήθελα να δράξω την ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για την ε, συνεργασιμότητά του και την συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου. Ε, ήθελα να, να, να σας επενέσω διότι πραγματικά ε, ε, ε, έχετε, οι, οι επιτυχίες οφείλονται σε εσάς Ο Βίκτορ είναι ικανοποιημένος. Ναι, όχι τόσο πολύ προσωπικά όσο για τα ωφέλη για τις περιφέρειες και είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς η Επιτροπή, πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η Επιτροπή, η Επιτροπή μας. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις θα προχωρήσουμε στη Ρίκα και την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Με την ευκαιρία του τελευταίου τριμερούς διαλόγου εξετάσαμε τα διάφορα άρθρα, το ένα δεν έχει πρόβλημα, μετά το 2021 και το 28. Για το 20 δεν υπάρχει επίσης πρόβλημα και συμφωνήσαμε και για το 21. Αποφασίσαμε λοιπόν όπως ξέρετε να δεχτούμε δύο τροπολογίες εδώ στο Κοινοβούλιο για να ενισχυθεί ο ρόλος αυτών των ευρωπαϊκών συσχε... συσσωματώσεων περιφερειακών μονάδων. Το 24α είναι στην αρρύθμιση του Συμβουλίου. Περί τίνος πρόκειται περί της συμμετοχής τρίτων χωρών σε αυτά τα προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο εξηγούν το ρόλο που πρέπει να παίζει αυτή η συνεργασία και αυτόν τον ρόλο τον συζητήσαμε πάρα πολύ. Και τελικά νομίζω ότι θα βρεθεί μια τεχνική λύση ώστε οι τρεις νομικές υπηρεσίες των τριών οργάνων να συνεννοηθούν Μόλις γίνει αυτή η συμβιβαστική πρόταση των νομικών υπηρεσιών θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Θα μπορέσουν να αρχίσουν. Η κοινοτική νομοθεσία θα είναι η βάση για την περιφερειακή αυτή συνεργασία από την οποία θα υποφεληθούν και τρίτες χώρες. Από την πλευρά των χωρών μελών αναφέρονται προβλήματα όπως η εθνική νομοθεσία που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων στις τρίτες χώρες. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι εθνικές νομοθεσίες και των χωρών αυτών. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν μπορεί να υπερισχύει πάντοτε και σε όλες τις περιπτώσεις επί της εθνικής εφόσον πρόκειται για τρίτες χώρες. Αλλά, αν κατάλαβα καλά, εμείς θελήσαμε γενικά να υπερισχύει η κοινοτική νομοθεσία. Πάντως και για τα τρία όργανα το σημαντικό είναι να καταλήξουμε σε μια λειτουργική αληθινή συνεργασία. Είναι τεχνικό το θέμα και είμαι σίγουρη ότι θα βρεθεί μια λύση και ένα συμβιβασμός. Και κάτι ακόμα. ακόμα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών την τελευταία φορά που συνεδρίασαν είπε ότι στον κανονισμό περιφερειακής συνεργασίας θα έπρεπε να αναφέρεται πολύ πιο συγκεκριμένα η συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Ξέρετε ότι στα πλαίσια του ΦΕΝΤΕΡ δίνεται αυτή η δυνατότητα συνεργασίας με τρίτες χώρες. Νομίζω όμως ότι κάτι παραπάνω πρέπει να γίνει μέσα στα πλαίσια αυτού του κανονισμού. Ίσως να το αναφέρουμε ήδη στο σκεπτικό ότι ενθαρρύνεται η συνεργασία και με τρίτες χώρες. Προβλέπεται τουλάχιστον. Εφόσον μάλιστα μπορεί να συνεισφέρουν και οικονομικά. Ο Καναδάς ενδιαφέρεται ας πούμε για τέτοια προγράμματα. Ελπίζω και από την Κομισιόν να έχουμε νέα και να υπάρξει συμφωνία για να μπορέσουμε όλα να τα λύσουμε. Να, αυτά για τον τριμερή διάλογο τον τελευταίο. Τη Δευτέρα νομίζω ότι θα ξαναβρεθούμε στον τριμερή διάλογο και τότε θα δούμε ποιες είναι οι επενδυτικές προτεραιότητες, άρθρα 5 και 6. Οι διαπραγματεύσεις θα είναι σκληρές νομίζω, αλλά πιστεύω επίσης ότι αν είμαστε ενωμένοι θα μπορέσουμε να υπερισχύσουμε και να συμφωνήσουμε και οι άλλοι. Λείπουν ακόμα, λείπει ακόμα συμφωνία για τα άρθρα 3 και 4, τη χρηματοδότηση δηλαδή. Και νομίζω ότι και εκεί θα περάσουν οι θέσεις μας. Το 7 έχει σχεδόν λυθεί. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια σύνδεση με το 87 του Γενικού Κανονισμού όπου ακόμα δεν έχουν λυθεί τα πάντα. Τώρα κάτι που δεν λύσαμε ακόμα είναι το θέμα των δικτών, αλλά αυτό είναι τεχνικό. Αυτά είναι, εκεί βρίσκεται η διαπραγμάτευση και νομίζω ότι σε λίγο θα καταλήξουμε σε συμφανία. Ευχαριστώ ακόμη μια φορά όλους τους διαπραγματευτάς. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση. Λάμπερτ. Ναι, ακούω ικανοποίηση με την πρόοδο, να σας συγχαρώ, αλλά αν θέλετε να πετύχετε όλα αυτά με τα μισά χρήματα, δεν θα είναι τόσο μεγάλη η ικανοποίηση. Πώς μπορείτε να συνεχίσετε με τον τρόπο αυτόν. μπορείτε να στείλετε σαφές μήνυμα ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν συνεχίσουμε έτσι. Δεν ε, θυμάμαι απ' έξω τα άρθρα που αναφέρατε, αλλά νομίζω ότι προσθέσατε μία προτεραιότητα, μία θεματική προτεραιότητα που θα επιλεγεί για, του, για τις συνοριακές περιοχές. Ε, αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό, διότι ο κύριος Χάνε σήμερα Μα ζήτησε να μην προσθέσουμε τίποτα, αλλά εμείς προσθέτουμε. Αν θυμάμαι καλά, στην θεματική συγκέντρωση ε, έχουμε μια ελεύθερη επιλογή για τις ε, ε, συνοριακές περιοχές. Τι γίνεται, το δεχτήκανε, πώς θα προχωρήσετε. Δεν έχουμε εξετάσει ακόμα τα άρθρα αυτά, τα άρθρα με τις προτεραιότητες αυτές. Θα επιμείνουμε όμως ε, και έχουμε πέντε επιλογές τις οποίες θα προτείνουμε αντί για τις τέσσερις που ε, περιέχονταν στην ε, πρόταση της Κομισιόν. Θα το διαπραγματευτούμε αυτό στο μέλλον όμως. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στο ερώτημα του Λάμπερτ. Πέρα από το ότι το Συμβούλιο προβλέπει ε, σκανδαλωδώς λίγα χρήματα για τις περιφέρειες, θα πρέπει να σκεφτούμε και εμείς πώς θα προχωρήσουμε, διότι συζητάμε τις τεχνικές λεπτομέρειες ε, που αφορούν όμως ε, και το θέμα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε και για νούμερα. Και μετά την απόφαση του, Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου της προηγούμενης εβδομάδας, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και κάποια στιγμή, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς πόσα χρήματα θα έχουμε για την περιφερειακή πολιτική, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν μας βοηθάει κανένα πλαίσιο. Εάν ε, δεν ε, μπορούμε να πετύχουμε κάποιους ε, δημοσιονομικούς πόρους. Και μετά από 36 ώρες διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο πιο πολλά ερωτήματα δημιουργεί παρά δίνει απαντήσεις. Τι γίνεται με τις επιστροφές για τις διάφορες περιφέρειες, τις εκτόσεις. Ε, πώς ε, θα συνυπολογιστούν αυτά με το συνολικό ποσό. Έχουν συμπεριλάβει πάρα πολλά σε μία απόφαση. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να μεταφερθούν αυτά στην πράξη και τι να σας πω, τρομάζω με την ιδέα. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε τι, πώς θα προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Ο Βίκτορ Ποστινάρου. Απλά να προσθέσω κάποιο δηλητήριο σε αυτή την ε, πολύ σκοτεινή εικόνα, γιατί έχουμε δύο κυρία θύματα των περικόπων προτείνονται από το είναι η εδαφική συνεργασία και το άλλο είναι το μέσιο διασύνδεσης της Ευρώπης, Connecting Group Facility. Τα κράτη-μέλη μη συνοχής ε, ε, ουσιαστικά από τους ε, είχαν εκτελεστεί ουσιαστικά από τους καθαρούς συνεισφέροντες. Τώρα όμως όταν βλέπουμε αυτά τα 20 εκατομμύρια, τα πρόσθετα 20 εκατομμύρια περικοπών ε, για τη συλλογή και για το Connecting Europe Facility, στην πράξη έχουμε δύο τρόπους με τους οποίους θα φυγούν οι, τις νεωρικές περιοχές. Δηλαδή, εκεί ξεκινά η ε, εδαφική συνεργασία και εκεί εμπλέκονται κοινότητες και θα είναι η μία συνέπεια εκεί και η δεύτερη συνέπεια θα είναι για το μέσο διασυνδέοντας την Ευρώπη και θα υπάρχουν συνέπειες γιατί οι κατανομές κονδυλίων ε, για στόχους όπως ε, θα είναι η ευρυζωνική διασύνδεση ή άλλοι στόχοι, δυστυχώς ε, δεν θα καλυφθούν. Ζήτω η στρατηγική του 2020 λοιπόν. Λοιπόν, Λάμπερτ. Αυτό που είπε ο κύριος Κέλλερ είναι σημαντικά. Δηλαδή, να δούμε πώς θα πράξουμε σαν επιτροπή, απευθείας όταν θα φτάσουμε στο κεφάλαιο αυτό, στο γενικό κανονισμό, σε αυτή τη χρηματοοικονομική παράγραφο ή ω ομάδε ή ω επιτροπή. Και θα έρθουμε σε επευθεία σε επικοινωνία με του διαπραγματευτές για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και κάθε φορά στο Στρασβούργο γίνεται μια συνάντηση για την ενημέρωση των συγκητών. Αυτό είναι σαφές. Ναι, Λαμασούρ, ξέρετε, πολύ, πολύ ξεκάθαρα στη Γαλλία, δεν μπορώ να το κάνω έτσι. Και είπε, ναι, περιορίσουμε, ας περιορίσουμε τον εαυτό μας ε, στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και όλα εμπίπτουν ε, στις ε, αρμοδιότητες των διαπραγματευτών. Και εγώ το ρώτησα, σίγουρος είσαι, γιατί αν δεν το αγγίξεις εσύ και το Συμβούλιο δεν μας ε, δώσει δυνατότητα να διαπραγματευτούμε. Όλα αυτά είναι ανοησίε. Εσύ πρέπει να αγωνιστεί για τα ίδια σημεία τα οποία αγωνιζόμαστε κι εμεί. Γιατί αν πει ότι δεν μα ενδιαφέρει το αποθυματικό επιδόσεων, τότε και το Συμβούλιο στην Κέσπη Διαπραγματεύση όχι είπε ότι αυτό είναι στο πακέτο του πολιτισμού συνομικού πλασίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε ποια είναι τα δικά μας κύρια θέματα και τι θα κάνουμε στα πλαίσια των δικών μας διαπραγματεύσεων, όμως τι θα πούν και οι κύριοι διαπραγματευτές για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί αν ε, ήταν ε, τόσο ξεκαθαρά τα πράγματα όπως είπε ο κ. δεν μπορούσα να συμφωνήσω, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος τελικά αν υπάρχει δυνατότητα ελιγμών. Ίσως να μπορούσε να μας βοηθήσει και ο Πρόεδρος και πάλι. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει να νιώθω παγιδευμένος. Lambert, when you are... Lambert. Φωνάζεις στη Ρίκα να αγωνιστεί εκείνη για τα χρήματα, αλλά η Κομισιόν είπε 11,6 δις, ο Φανρόμπε είπε 8,9. Τώρα λοιπόν εμείς πρέπει να αποφασίσουμε να βάλουμε ένα ποσό στο νομοθετικό πλαίσιο και να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Ο Πίτερ νομίζω κάτι ήθελε να πει. Το ίδιο θέλω να πω. Αυτό που μόλις είπες, ότι και στον γενικό κανονισμό στο 8,4 στο 8,4 συμπεριλαμβάνεται αυτό. Ε, είναι πολύ σημαντικό ε, και από τι δύο πλευρέ η Κομισιόν είπε ότι χρειαζόμαστε περισσότερου πόρου στο θέμα αυτό. Ήθελα να πω κάτι για τα εξωτερικά σύνορα. Ήταν σημαντικό θέμα ε, συνεργασίας ε, στην παρούσα περίοδο, ήταν όμω και δύσκολο. Έχουμε την αίσθηση ότι το συμβαστικό κείμενο που επιτεύχθη είναι σημαντικό βήμα προόδου. Απέτησε πολλή δουλειά και από τα τρία θεσμικά όργανα και από τις νομικές υπηρεσίες. Νομίζω όμως ότι τώρα πια έχουμε ένα κείμενο το οποίο θα ε, ε, δώσει περισσότερη σαφήνεια στο μέλλον και όπως είπε ο εισηγητής ε, είμαστε διατεθειμένοι να δούμε πώς μπορούμε να διασαφηνίσουμε την πτυχή αυτή στον κανονισμό. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλεις να ξαναπάρεις το λόγο. Ε, Όσον αφορά τις παρατηρήσεις μας ε, για τον ε, προϋπολογισμό, ως ε, Κοινοβούλιο θα πρέπει να αγωνιστούμε για να, έχουμε, για να πετύχουμε περισσότερους πόρους για την περιφερειακή συνεργασία, αλλά έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Και το Συμβούλιο είπε ότι θα πρέπει να πούμε από πού θα ληφθούν τα χρήματα εάν θέλουμε περισσότερα. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή μας να δει ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Και οι συνάδελφοι ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα στις πολιτικές τους ομάδες. Ε, καλό θα ήταν εάν μπορούμε να λάβουμε απόφαση πριν ε, ψηφίσουμε για το δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά συμφωνήσαμε ότι δεν θα συζητήσουμε νούμερα, γι' αυτό δεν θίξαμε αυτό το ερώτημα, αλλά όπως είπε ο Βίκτορ, είναι ακατανόητο το Συμβούλιο να κάνει περικοπές ακριβώς στο θέμα της ε, περιφερειακής συνεργασίας που αποτελεί τη βάση της καλής ευρωπαϊκής συνεργασίας. Ελπίζω να συνεχιστούν οι συζητήσεις ε, και να Είμαστε ε, δραστήριοι και στον γενικό κανονισμό ώστε να αγωνιστούμε ε, για το θέμα αυτό, διότι έχουμε σαφή εντολή και όσον αφορά την ε, θεματική συγκέντρωση που ανέφερε, συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 5. Σίγουρα λοιπόν θα το συζητήσουμε αυτό στην επόμενη μα συνεδρίαση. Ευχαριστώ και για το τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ε, ναι, έχουμε τον ε, κανονισμό για την ε, εδαφική συνεργασία. Δεν είναι νέος, είναι τροποποιημένος όμως βασίζεται στον ισχύοντα, είναι νομικό μέσο, δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με χρήμα ή με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι ένα ιδιαίτερο θέμα, δεν είναι ιδιαίτερα ογκώδης ο κανονισμός αυτός. Ωστόσο υπάρχουν και εδώ κάποια ε, σημαντικά θέματα. Όπως έχω ήδη ε, πει, ε, είμαι γνώμων προς την Ιρλανδική Προεδρία που έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, διότι η προηγούμενη Προεδρία δεν ασχολήθηκε. Στις 4 Μαρτίου λοιπόν είχαμε την πρώτη διαπραγμάτευση σε τριμερή διάλογο όπου προείδευσε η πρόεδρος της Επιτροπής μας ε, και μπορέσαμε να πετύχουμε ήδη κάποια πράγματα. Το θέμα λοιπόν είναι... Ε, τι θέλουμε λοιπόν, ε, αποσαφήνιση, απλούστευση και βελτίωση της διαδικασίας ε, ίδρυσης και εφαρμογής των ομίλων. Ε, η συνάδελφος Ερίκα Μάνερ αναφέρθηκε στο θέμα ε, δημιουργίας ομίλων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Συμφωνία μπορούσε ήδη να επιτευχθεί όσον αφορά το ε, εφαρμοστέο δίκαιο ε, και την ρήτρα που αφορά τη Λισαβόνα. Ε, είναι σαφές λοιπόν το θέμα αυτό. Αυτό που δεν είναι ακόμα απόλυτα σαφές είναι αυτό που ανέφερε η Ρίκα Μάνερ. Το εφαρμοστέο δίκαιο για τους ομίλους εδαφικής συνεργασίας ε, που θα ιδρύονται μαζί με ε, περιφέρειες από τρίτες χώρες, διότι αυτό άπτεται και τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής. Ψάχνουμε λοιπόν για σχετικές λύσεις. Επίσης, ε, συζητήσαμε το θέμα της ε, αδειοδότησης, της έγκρισης. Υπάρχουν λοιπόν εδώ κάποια θέματα στα οποία θα μπορέσουμε να βρούμε συμφωνία, την οποία δεν έχουμε βρει ακόμα. Ε, έχουμε, συζητήσει, έχουμε και το θέμα της προσχώρησης νέων μελών σε ήδη υπάρχοντες ομίλους. Άλλα θέματα είναι η συμμετοχή τρίτων χωρών, η ε, συμμετοχή δημοσίων φορέων και ομιλή εδαφικής ε, συνεργασίας ε, και διαχείριση του προσωπικού. Επίσης θέμα ευθύνης των ομίλων αυτών. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε με την Προεδρία του Συμβουλίου την επόμενη Πέμπτη. Στο μεταξύ έχουμε πάνω από 30 τέτοιους ομίλους. Ε, πολλές ε, περιφέρειες σκέφτονται τη δημιουργία τέτοιου ομίλου, περιμένουν όμως τον νέο κανονισμό. Υπάρχουν ε, ακόμα προβλήματα διοικητικά όσον αφορά τη διαχείριση του προσωπικού και βασικός μας στόχος είναι να ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια για τους υπάρχοντες και τους νέους ομίλους. Αυτό είναι το... Αυτά λέει η εντολή που έχω λάβει από την Επιτροπή μας. Ε, σημαντικό είναι να διατηρήσουμε τις προτεραιότητες που έχουμε στον τριμερή διάλογο. Ε, σημαντικό θέμα είναι η... Ε, η ε, αδειοδότηση με, τις, ε, με τη διαδικασία της ε, σιωπή. Κάτι τέτοιο είχε συμπεριληφθεί στην πρόταση της Κομισιόν. Εμείς είμαστε θετικοί απέναντι. Σε αυτό προβλέπεται εξάμεινη προθεσμία μετά την υποβολή της αίτησης. Στόχος είναι να αποφύγουμε διακοπή αυτής της προθεσμίας στα αγγλικά είναι Tacent Approval ε, και θα πρέπει να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Ε, το Συμβούλιο προτείνει παρέκκληση για τα κράτη-μέλη στα οποία έχει την έδρα του ο μελλοντικός όμιλος. Αυτό όμως θα υπονομεύσει τον νόμο διότι το, στο παρελθόν είδαμε ότι ειδικά αυτά τα κράτη-μέλη ε, είχαν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις ε, κατά τη διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν να διαπραγματευτούμε το θέμα αυτό. Επίσης ε, επιμένουμε σύμφωνα με την συμφωνούμε με, σύμφωνα με την ε, εντολή μας επιμένουμε ε, στο θέμα του ε, εισοδήματος και όχι της επένδυσης στον όμιλο. Πιστεύουμε ότι η αλλαγή του κανόνα αυτού θα επιφέρει σημαντικό γραφειοκρατικό άχθος και η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου βρίσκεται στο πλευρό μας, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει αντίθεση από διάφορα κράτη-μέλη. Δεύτερο σημαντικό θέμα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο εργασίας, το εφαρμοστέο εργασιακό δίκαιο. Ε, οι όμιλοι αυτοί χρειάζονται ευέλικτους αλλά σαφείς κανόνες ε, για την ε, πρόσληψη και διαχείριση του προσωπικού για να αποφύγουμε κατακαιρματισμό των κανόνων και μη διαφανείς κανόνες. Διότι κάτι τέτοιο θα έχει ανεπιθύμητες ενέργειες για το προσωπικό που εργάζεται σε έναν Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας. Η ε, δυνατότητα επιλογής ε, που προτείνεται από την Κομισιόν θα επιφέρει την ε, επιθυμητή ευελιξία Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα έχουμε επιθύμητα αποτελέσματα. αλλά υπάρχουν κράτη-μέλη που διαφωνούν με αυτό, αλλά και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Επίσης έχουμε την ε, συμμετοχή των τρίτων ε, χωρών. Στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων ε, θα θέλουμε απλοποίηση και διασαφήνιση σχετικά με τη συμμετοχή των τρίτων χωρών. Κάποια κράτη-μέλη θέλουν να διατηρήσουν τη δυνατότητα για τις υπερπόντιες περιοχές τους. Ήδη Έχουμε το μέσο γειτονίας, ε, το μέσο προσχώρησης. Ναι. Σε άλλες επιτροπές, όπως την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων, συζητώνται τα θέματα αυτά όπως και η δυνατότητα συνεργασίας ε, περιφερειακών, ε, ε, συνοριακών περιοχών με βάση έναν Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας. δεν είναι επίμαχο λοιπόν το θέμα της ε, συμμετοχής των τρίτων χωρών, το θέμα είναι ποια νομική βάση θα επιλεγεί. Ε, άλλο θέμα που εκκρεμεί είναι η συμμετοχή δημοσίων φορέων. Εμείς επιμένουμε ότι κάτι τέτοιο θα είναι ε, σημαντική είναι απαραίτητη όμως σε τομείς όπως είναι οι μεταφορές, η υγεία, η ε, παροχή νερού κλπ. Έτσι θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τους τομείς αυτούς. Και τέλος, το πέμπτο σημαντικό σύμπλεγμα που θα πρέπει να διαπραγματευτούμε είναι η τομεακή πολιτική και η συμμετοχή ε, σε δημόσιους διαγωνισμούς. Ε, οι όμιλοι αυτοί θα πρέπει να έχουν πιο σημαντική θέση στο μέλλον ε, στις ε, τομεακές πολιτικές και θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς. Αυτά λοιπόν ήταν τα πέντε σημαντικά συμπλέγματα προβλημάτων το οποίο θα πρέπει να διαπραγματευτούμε. Την Πέμπτη θα συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις και για τον Απρίλιο ήδη έχουμε ορίσει κάποιες ημερομηνίες. Η Ιρλανδική Προεδρία έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ε, μέχρι το καλοκαίρι. Ε, η Ιρλανδική Προεδρία είναι αρκετά συνεργάσιμη, κάποια κράτη-μέλη αντιτίθενται, ειδικά αυτά με, κεντρική, με σημαντική κεντρική διοίκηση. Θα πρέπει όμως πιστεύουμε να ε, ε χαλαρώσουν κάπως τη θέση τους αυτά τα κράτη-μέλη. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει κανένα άλλο σχόλιο. Όχι. Ραμπέ ούτε λίγο. Α, ούτε λίγο. Καλά, εντάξει. εντάξει, αλλά μην προλέγουμε κιόλα, λοιπόν. Ευχαριστούμε Ιωακήμ. Δεν σε εμπόδισε κανείς νομίζω από άλλες ομάδες οπότε μπορείς να κινηθείς. Εδώ λίγη συνεδρίαση. Θα ξαναβρεθούμε για δύο μισές μέρες τον Απρίλιο. Αυτά ευχαριστώ τους πάντες και τους διερμηνείς. Ευχαριστώ φύγετε τώρα.